Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Η ημερησία μας διάταξη είναι πάρα πολύ βεβαιωμένη. Η συνεδρίαση είναι πολύ σύντομη και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κατά το μέγιστο το χρόνο μα. Θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία μεταξύ ημών του Προέδρου Μέντστατ και του Μισελ Πλουνσού το Γενικό Διευθυντικό του ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που του ανατέθηκε από το Συμβούλιο μία έρευνα για τι εξωτερικέ ασχέσει τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεω, σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη, και που είναι ήδη παρόν από την αρχή των εργασιών μα. Περιμένοντα τη συζήτηση του σημείου 4. Όσον αφορά το σημείο 1, είδατε το σχέδιο σημείο της διάταξης, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται. Θα υπάρχουν μικρές αλλαγές, όχι στο περιεχόμενο, αλλά στη σειρά των σημείων. Ιδίω η, ε, η, κυρία Χάουκ ζήτησε το σημείο 18 να εξαρθεί μετά το σημείο 6. Και το σημείο 7 με εξεταστεί μετά το 17. Ο Γενικό Γραμματέα ο Σεβλέ ζήτησε να είναι παρόν στη συζήτηση αυτή για να απαντήσει σε ενδεχόμενε ερωτήσει. Έχει απόλυτο δικαίωμα να το κάνει. Θα το ξέρουμε λοιπόν στι 6 4, παρά 20. Έχετε το κατάλογο των διαθεσίμων του Χιλόσο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όπως όλες μας συνεδριάσεις και αυτή αναμεταδίδεται άμεσα στη σωσίδια του Κοινοβουλίου και θα ήθελα από την άλλη μεριά να σας πω επίσης ότι από τους συνεργάτες μας χάνουμε την Βίρτο Κόικα που θα φύγει από τη γραμματεία η διορίστηκε επικεφαλή τη υπηρεσία Ιντερνετ, στη Γενική Διευθυνσία Ιντερνετ. Την συγχαίρουμε και εκφράζουμε βέβαια τη λύπη μας για την ενοχώρησή τη. Ε, merci pour elle. En point 3, approbation euh, des... Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων. 20 Ιανουαρίου και 26 Ιανουαρίου. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά αυτά ενεκρίθησαν. Περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 4 που αφορά τα συμπεράσματα και συστάσεις της ε, εντολής που δόθηκε στον κύριο Καμπτεσί για τις εξωτερικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πρόκειται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα να σας πω ότι πρότεινα τους άλλους προέδρους των ε, εμπλεκομένων επιτροπών, στις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δηλαδή, να έρθουν εδώ. Και θα έχουμε έτσι συμμετοχή του κυρίου Ντότς, που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προπολογισμού και είναι και εισηγητής για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη δική Επιτροπή, εξ ονόματος της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, την κυρία Γκιορή επίσης εισηγήτρια, και εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης, τον κύριο Μπέρμαν, επίση εισηγητή για το ίδιο θέμα. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εξωτερικού Εμπορίου δυστυχώ δεν μπόρεσαν να αποστείλουν κάποιον να του εκπροσωπεύσει. Πριν δώσω το λίγο στον κύριο Καμτεσού, η κυρία Καβάλα και ο κύριο Φερνάν ζήτησαν για διαδικαστικό θέμα το λόγο. Παρακαλώ. Eh, um Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σα μιλήσω για ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε, την κατάσταση στη Μαδέρα. Ξέρετε ότι η Μαδέρα καταστράφηκε πραγματικά από μια θεομηνία ο αριθμός ε, των νεκρών και των τραυματιών είναι εξαιρετικά υψηλός, ενώ οι υλικέ ζημιές εξίσου σημαντικές, ιδίω σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την ίδρυυση. Η, το νησί, η Μαδέρα νομίζω ότι χρειάζεται την ελεγγύη μας. Όλοι οι Πορτογάλοι βουλευτές του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούν να οργανώσουν μια κοινή δράση θα υποβάλουν κάποιες προτάσεις σχετικά αύριο και είμαι πεπισμένη ότι η κυβέρνηση ότι θα υπάρξει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά να σας ενημερώσω ότι θα υποβληθεί επίσημο αίτημα προς την, Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ από τους συναδέλφους την αλληλεγγύη στην Μαδέρα. Ευχαριστώ συνάδελφε πραγματικά μας συγκλώνησε όλους η τραγωδία στη Μαδέρα και οι εικόνες που είδαμε στην τηλεόραση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσε την πρότασή σας, είμαι πεπισμένος ότι όλα τα όργανα της Ένωσης επιθυμούν να υλοποιήσουν τις διαδικασίε που διαθέτουν και να χρησιμοποιήσουν την υφισταμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσουν τον πληθυσμό του νησιού. Η κυρία Ζολή, πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, ήρθε και αυτή, την καλωσορίζουμε. Δίνω το λόγο στον Μισελ Καμτσού. Υπενθυμίζω ότι τον ζητάνε από παντού. Είναι μεταξύ των σοφών που όλοι οι διεθνείς οργανισμοί επιδιώκουν να ε, καλέσουν και να συμπεριλάβουν για να εκμεταλλευτούν την με μεγάλη εμπειρία που έχει στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά σε διεθνές επίπεδο. Το Συμβούλιο ιδίω θέλησε να ακούσει την ανάλυση και τις συστάσεις του για το ρόλο της ΕΤΕΠ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης στο ενδιάμεσο της περιοδου 2007-2013. συζητώντα με τον πρόεδρο κύριο Μετσά, τον κύριο Καμψίου και εμένα, σκεφτήκαμε, και εγώ σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον μετά την κατάθεση τη έκθεση στον πρόεδρο των, στους πρόεδρους των θεσμικών οργάνων να έρθει εδώ ο κύριος Καμπτεσού για να μας ενημερώσει για τα συμπεράσματα και να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων που θα βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τις εργασίες για την αναθεώρηση και την ενδιάμεση εξέταση της ε, δραστηριότητες ΕΤΕΠ που μπορεί να γίνει πραγματικά βασικό εργαλείο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας δίνω το λόγο αγαπητέ φίλε και σας ευχαριστώ ξανά που δεχθήκατε να, παραστεί, να παρουσιαστείτε ενώπιόν μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας πω καταρχήν ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να λαμβάνω το λόγο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πίστευω ότι θα είχα ποτέ μια τέτοια τιμή στη ζωή μου. Το λέω αυτό πραγματικά, αλλά αυτό το απολαμβάνω ακόμη περισσότερο. Όντως, μου ανατέθηκε η Προεδρία της Επιτροπής Σοφών που αναφέρατε. Ήταν δέκα οι σοφοί και εγώ είχαμε κληθεί όλοι να εξετάσουμε εν μέση οδό, όπως λένε, την, τον τρόπο υλοποίησης της σημαντικής εντολής που είχε ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων του 2007. Η... Κάναμε αυτή τη δουλειά το 2008 και 2009 εξετάζοντας την κατάσταση ως λεπτομεριακοί εξωτερικοί αξιολογητές, βλέποντας τι έγινε και τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Και μπορώ να σας πω ότι παρότι η ΕΤΕΠ δουλεύει πάρα πολύ καλά, υπάρχουν ακόμα πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ο κόσμος άλλαξε. Και η Ευρώπη και μάλιστα άλλαξαν ριζικά. Notre groupe, euh, non sans quelques hésitations, a pensé que είχαμε κάποιους δισταγμούς στην ομάδα, αλλά θεωρήσαμε εν τέλει ότι δεν θα ήταν σωστή η απάντηση στην εμπιστοσύνη που μας είχε δοθεί αν μέναμε σε μια ε, κυριολεκτική και περιοριστική ανάλυση της εντολής και εξετάζαμε μόνο τι λειτουργούσε, τι δεν λειτουργούσε καλά. Θέλαμε να προβλέψουμε τον επερχόμενο πόλεμο όπως κάνουμε μερικές φορές η στρατηγοί, όχι απλά να πολεμήσουμε τον υφιστάμενο. Θέλαμε να δούμε τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε στην ΕΤΕΠ μετά από αυτή την κρίση που συγκλώνησε, που ανατάραξε τον κόσμο, μετά την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, μετά την ε, συνένεση που υπήρξε ε, μεταξύ Κοινοβουλίου Συμβουλίου για τα θέματα της αναπτυξιακής πολιτικής. Μια σειρά αλλαγών υπήρξαν, δεν θέλω να τις αναφέρω όλες, που μας στο να πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε τι χρειαζόταν να γίνει στην τράπεζα, γιατί η κατάσταση στο μέλλον ε, θα ήταν πολύ διαφορετική και δεν θέλαμε να θεωρήσουμε ότι ο κόσμος λύγει το 2013 και δεν αλλάζει ποτέ ξανά τίποτα. Ως εκ τούτου επειδή όμως η εντολή μας ήταν διαφορετική, την, την εισήγησή μας την κάναμε σε δύο τμήματα. Πρώτον, η υφιστάμενη κατάσταση με συγκεκριμένες συστάσεις και ένα δεύτερο τμήμα όπου με κάποιο κάπως παράτολμα προσπαθούσαμε να διερευνήσουμε τι θα μπορούσε να γίνει η ΕΤΕΠ μετά το 2014 μέχρι το 2020 ενδεχόμενα για να εξυπηρετήσει καλύτερα τις φιλοδοξίες της Ευρώπης ιδίως στο πλαίσιο τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι σαφές ότι υπάρχει μία ενεργή παρουσία της Ευρώπης, οικονομικού χαρακτήρα και αναπτυξιακού χαρακτήρα, πέραν των διπλωματικών αποστολών και ότι μπορεί να γίνει ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο πρωταρχικό προτείνοντας μια σειρά επιλογών, δύο επιλογές, που θα, από τις οποίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη μελέτη τους οι κυβερνήσεις. Ας μιλήσουμε πρώτα για τις συστάσεις για το άμεσο μέλλον. Ξεκινώ με μια παρατήρηση. Δεν θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι διαπιστώσαμε πως η ΕΤΕΠ έστω και αν την συγκρίνουμε με, άλλα διεθνή, με άλλους διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που εξυπηρετεί την Ένωση. Και θέλω να το πω αυτό παρόντος του κ. Μεϊστάτ. Είναι αποτελεσματική, ικανή, προσφέρει προς τη θέμενη αξία μεγάλη στα πλαίσια των ορίων που της έχει θέσει το καταστατικό της. Σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές της δραστηριότητες, που αποτελούν μόνο το 10% των συνολικών δραστηριοτήτων της, σιγά σιγά και σχεδόν κρυφά έγινε ένα πρωταρχικό εργαλείο αναπτυξιακή πολιτική. Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμο εύκολα. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πακέτο εξωτερικέ δράσει έχει το ίδιο μέγεθο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικονόμηση και την Ανάπτυξη, η τράπεζα Ιμπέρντ στο Λονδίνο και είναι, έχει διπλό μέγεθο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανάπτυξη, ενώ είναι το ίμιση τη Παγκόσμια Τράπεζα χοντρικά. Αυτό αφορά μόνο το εξωτερικό της πακέτο. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από την Παγκόσμια Τράπεζα αν πέραμε και το εσωτερικό και την εσωτερική, τη διάσταση εσωτερικών πολιτικών. Άρα γίνεται ένα πρωταρχικό εργαλείο προς όφελο της Ένωσης. Και προσθέτω την άποψη της ομάδας μας ότι δεν έχει φτάσει στα όρια τη το επίπεδο αυτό. Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερο για να εξυπηρετήσει τις ευρωπαϊκές επιθυμίες εφόσον βεβαίως προσαρμοστεί στην εντολή εφόσον προσαρμοστούν οι πόροι πάντως μπορεί να δώσει περισσότερα αποτελέσματα. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Και αυτό μας το παρατήρησαν οι εξωτερικοί αξιολογητές. Η τράπεζα είναι τρόπον Α εν κάπως θύμα της αρετής της. Είναι μία τράπεζα που είναι εξαιρετικά επιφυλακτική και όταν ε, τίθεται ζήτημα αύξησης του προσωπικού της. Σε τέτοιο βαθμό που θα δείτε και στην έκθεση σελίδα 62 περιλαμβάνεται εκεί κάτι εξαιρετικά εύγλωτο. Στην ΕΤΕΠ υπάρχουν πολύ λιγότεροι υπάλληλοι ανά χορηγηθέν δάνειο από άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στις ικανότητες του κύριου Μεϊστάτ, αλλά και διότι στις εξωτερικές της δράσεις εφάρμοσε τις ίδιες μεθόδους και τα ίδια περιορισμένα μέσα που εφαρμόζει στις δραστηριότητές της του της Ένωσης. Εδώ όμως ανακύπτει το πρόβλημα. Εάν θέλουμε, όπως η συνένεση που υιοθετήσετε το απαιτεί, να της δώσουμε έναν ρόλο χρηματοδότη της ανάπτυξης, που είναι, και σας λέω μια προσωπική μου άποψη, μια καλή ιδέα, τότε είναι σαφές ότι θα έπρεπε να αναβαθμιστούν τα υλικά της μέσα. Δεν δανείζεις με τον ίδιο τρόπο μια χώρα της Ένωσης και με τον ίδιο τρόπο μια χώρα που έχει πολύ μικρότερη θεσμική υποστήριξη, όπου χρειάζεται μεγαλύτερη παρακολούθηση των έργων, πολύ λεπτομερίστερη εξέταση των προτάσεων κλπ. Άρα η κυρίαρχη παρατήρηση της ομάδας μας είναι ότι η τράπεζα μπορεί να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά προς όφελος της Ένωσης εάν ξέρουμε και εσείς εάν αποφασίσουμε και εσείς το αποφασίσετε να τις τα ανθρώπινα και οργανωτικά μέσα που είναι αναγκαία για να κάνει τη δουλειά της. Αυτή είναι η πιο γενική παρατήρηση. Πέραν αυτών η ομάδα έχει έξι βασικές ε, συστάσεις. Πρώτον, και αυτό είναι δική σας δουλειά γιατί εσείς συναποφασίζετε με το Συμβούλιο. Ε, μιλώ για την ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού και υλοποίηση της εντολή, των εντολών αυτών. Εμείς πιστεύουμε ότι τα θέματα που εμπεριέχει η εντολή είναι τα ενδεδειγμένα. Οικονομικές υποδομές, ε, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, χρηματοδότηση και υποστήριξη επενδύσεων ε, ιδιωτικού χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο, υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι στόχοι που εσείς θεωρείτε στόχου στόχους προτεραιότητες ανά περιφέρεια δεν δημιουργούν πρόβλημα. Ωστόσο είναι καθοριστικό το Κοινοβούλιο να συνεχίζει να καθορίζει τους στόχους προτεραιότητας, δράσης προτεραιότητας της ΕΤΕΠ και τα οικονομικά πακέτα για κάθε ε, κατεύθυνση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι νωρίτερα. Να φροντίσουμε δηλαδή ώστε ο συντονισμός μεταξύ Επιτροπής και Τράπεζας να είναι πιο, πιο στενός όταν θέλουμε να καθορίσουμε συγκεκριμένα ε, επιχειρησιακούς προσανατολισμούς. Εδώ χρειάζεται μια σειρά συντονιστικών, ε, συντονιστικού χαρακτήρα επικοινωνιών μεταξύ τράπεζας και επιτροπής, ούτως ώστε οι προτεραιότητες που εσείς υιοθετείτε να υλοποιούνται με πιο συγκεκριμένο τρόπο και να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις επιχειρησιακές αποφάσεις. Επίσης, μια άλλη παρατήρησή μας, σε έναν τόσο μεταβαλλόμενο κόσμο, το να θέτουμε στόχους για 7 χρόνια γίνεται ίσως υπερβολικά φιλόδοξο. Θα πρέπει να προσφέρουμε τη δυνατότητα στην τράπεζα να αλλάζει πορεία καθοδόν το Συστήνουμε λοιπόν να υπάρχει μια κάποια ευελιξία εδώ. Μετά την πρώτη αυτή προχωρούμε σε μια δεύτερη σύσταση που δίνει συνέχεια στη συνένεση που εγκρίνεται σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Πιστεύουμε ότι, και εσείς το είπατε, ότι η, τράπεζα δέχεται να αλλάξει στον τομέα και να γίνει κάτι που δεν είναι. Μία τράπεζα που θα χορηγεί ενισχύσει αναπτυξιακού χαρακτήρα. Μην ξεχνάτε ότι η ΕΤΕΠ ε, είχε ε, επινοηθεί ω τράπεζα ε, ενίσχυση των επενδύσεων. Αυτή ήταν η αρχική τη ιδέα. Τώρα πρέπει να ξεπεράσει ένα πολύ σημαντικό βήμα, να γίνει δηλαδή μια τράπεζα που υποστηρίζει και την ανάπτυξη. Πρέπει να ξέρουμε ωστόσο ότι τούτο δεν γίνεται εν μία ανοιχτή. Ούτε με ένα τσακ. Πρέπει να αλλάξουν όχι μόνο τα μέσα ε, βαθιά, αλλά να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο και η κουλτούρα της τράπεζας. Αυτό απαιτεί χρόνο, σας το λέω με βεβαιότητα. Τόσο ο πρόεδρος όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θέλουν να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, αυτό θα γίνει πραγματικότητα μόνο αν επιτρέψουμε στην τράπεζα να προσλάβει ανθρώπους για να διαχειριστούν τέτοιες πολιτικές και αν στις σχέσεις της με την Επιτροπή υπάρχουν διαδικασίες blending, δηλαδή της ε, ανάμιξης δωρεών και δανείων. Αυτό θα πάρει χρόνο, προφανώς. Βραχυπρόθεσμα ωστόσο η τράπεζα θα πρέπει να προσέξει ακόμα περισσότερο θέματα που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη, όπως η αλλαγή του κλίματος και η προσαρμογή των χωρών στις αλλαγές του κλίματος, με ό,τι περιλαμβάνει αυτό σε χορήγηση δωρεάς πέραν των δανείων. Να δίνει έμφαση στις τοπικές επενδύσεις και τις υποδομές που έχουν αντίκτυπο στην αναπτυξιακή πολιτική, να ενισχύσει την προσοχή της στα κοινωνικά θέματα, σε ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε ζητήματα που σχετίζονται με την πρόληψη ή την, επίληψη, την επίλυση συγγνώμη, σειράξεων. Όλα αυτά είναι τμήμα της συνένεσης για την ανάπτυξη. Πρέπει να υλοποιηθούν από την τράπεζα, να γίνουν και με μια προσέγγιση προοδευτική ανάμεσα, ανάλογα και με, τις, ε, τα μέσα που θα διαθέτει. Ένα τρίτο ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μία απόφαση που πρέπει να ληφθεί για το αν τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία υφίστανται ως εθελούσια εντολή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ή αν θα πρέπει να ακυρωθεί η δυνατότητα αυτή. Η δική μας ομάδα πιστεύει ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν τα κονδύλια αυτά και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επιτόπου βέβαια με δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τα περιφερειακά κονδύλια τα οποία έχετε εσείς καθορίσει, δίνοντας περισσότερα στις ε, χώρες, ε, της υποψήφιες ή στις ε, όμορες μας χώρες. Πιστεύουμε ότι η κατανομή των περιφερειακών κονδυλίων έχει γίνει σωστά. Πιστεύουμε πάντως ότι μετά από τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία δεν θα έλεγα ότι είναι αποτελέσματα της Κοπενχάγης, είναι πάντως πολύ σημαντικό να αυξήσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών και για την προσαρμογή των χωρών που πλήττονται από τα φαινόμενα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο σας προτείνουμε να χορηγήσετε το ποσό αυτό κυρίως για τα ζητήματα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Αλλά αυτό θα γίνει, όπως σας είπαμε, δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να δημιουργήσουμε την κατάλληλη και αποτελεσματική ανάμιξη δωρεών και δανείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτον λοιπόν αυτών και από την άλλη στη χορήγηση των δανείων αυτών όλες οι συστάσεις που κάνουμε για καλύτερο συντονισμό, για καλύτερη αποτελεσματικότητα της ε, συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να ε, τηρηθεί σε κάθε περίπτωση. Και έπειτα τρίτο ή τέταρτο σημείο στις συστάσεις μου μας ε, ζητήθηκε να δούμε αν υπήρχε ένα, ένας τρόπος να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία, ακόμα και αν υφίσταται ήδη αυτή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο ακολουθεί. Πολύ σύντομα θα, να σας πω το εξή: Όπως και στον αθλητισμό δεν αλλάζουμε μια ομάδα η οποία κερδίζει έτσι και στις δικές μας εργασίες δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να αλλάξουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Ωστόσο όμως, ακριβώς επειδή πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερους πόρους, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και περισσότερο την εγγύηση, την κοινοτική εγγύηση που δίδεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θεωρούμε ότι πολλές επιχειρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή με την εγγύηση, στα πλαίσια της εγγύησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαν να γίνουν, ε, δεδομένων της πρόοδου που έχει σημειωθεί σε διάφορες χώρες, θα μπορούσαν λοιπόν να γίνουν ε, με ίδιο κίνδυνο της τράπεζας πράγμα το οποίο θα μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε άλλες δράσεις που να καλύπτονται από την κοινοτική εγγύηση. Σας ε, ζητώ λοιπόν να, γίνει ένα graduation, όπως τα λέγαμε στα αγγλικά, των δραστηριοτήτων, μια διαβάθμιση των δραστηριοτήτων της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προκειμένου να καταφέρουμε να περάσουμε κάποιες δραστηριότητές μας ε, στα πλαίσια ανάληψης ιδίου κινδύνου της τράπεζας, χωρίς να καλύπτονται οι δράσεις αυτές απαραίτητα από την κοινοτική εγγύηση. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο δράσεις τεχνικής αρρωγής προς αναπτυσσόμενες χώρες, δράσεις για την ισχυροποίηση του θεσμικού πλαισίου στις χώρες αυτές και νομίζω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τις πολιτικές ανάπτυξης. Μέχρι στιγμή οι περισσότερε αυτέ δράσει γινόντουσαν με χρηματοδότηση από του κοινοτικού πόρου, από του πόρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι ένα μέρο των δραστηριοτήτων αυτών θα μπορούσε να γίνουν με του ίδιου πόρου τη ΕΤΕΠ. Αυτή λοιπόν είναι μία από τι συστάσει μα που μπορείτε να δείτε στην έκθεσή μα. Επίση, πολλά πράγματα θα μπορούσε να πει κανεί για τη συνεργασία με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, κυρίω τα πολυμερή χρηματοοικονομικά θεσμικά όργανα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δείτε ότι η έκθεσή μας κάνει πάρα πολλές σχετικές συστάσεις και μπορώ να σας πω ότι ε, και από τις δύο πλευρές υπάρχει μια πολύ καλή βούληση για να κατευθυνθούμε προς την ε, κατεύθυνση αυτή, ιδίω όσον αφορά τις δράσεις αυτές που, ε, στις οποίες ζητάμε να γίνει μια καλή ανάμειξη δωρεών και δανείων. Η συνεργασία λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει για τις προτάσεις αυτές, ενδεχομένω όχι με τους γρήγορους ρυθμούς που θα προτιμούσαμε, αλλά έχει ξεκινήσει τουλάχιστον η συνεργασία. Βέβαια, ένα δύσκολο ζήτημα της διεθνούς συνεργασίας, και εδώ πέρα αναφέρομαι και στο ένοχο παρελθόν, αν θέλετε, είναι η συνεργασία μεταξύ των πολυμερών χρηματοοικονομικών οργανισμών. στις συνεδριάσεις του G7, του G8, του G... ό,τι θέλετε ουσιαστικά. Πολλές φορές αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να συντονιστούν καλύτεροι οργανισμοί. Και το λέμε αυτό κυρίως όταν δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο να πούμε. Καλούμε λοιπόν τους οργανισμούς αυτούς να συνεργαστούν περισσότερο, να συντονιστούν περισσότερο. Θα έλεγα ότι η ρήτρα αυτή, μόλον ότι ακούγεται κάπως επιθετική, τελικά είναι χρήσιμη, γιατί όντω τελικά συμβάλλει στο να βελτιωθούν τα πράγματα. Αλλά όπως το ξέρετε, τα θεσμικά όργανα είναι τελικά θεσμικά όργανα και κάθε θεσμικό όργανο, κάθε οργανισμός οχυρώνεται στο δικό του πλαίσιο και έχει βέβαια σωστούς λόγους κάθε οργανισμός για να κάνει κάτι τέτοιο. Του ζητάμε βέβαια να συνεργαστούν όλο και περισσότερο. Βρισκόμαστε λοιπόν, αν θέλετε, στην μαύρη αυτή τρύπα της διεθνούς συνεργασίας, όπου καλούμεθα κάθε φορά να σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο, υπάρχουν σαφώς περιθώρια βελτίωσης, αλλά υπάρχει και ένα γυάλι, μια γυάλινη οροφή την οποία δεν μπορούμε να περάσουμε αν δεν αλλάξουμε κάπως την ε, οριοθέτηση των ε, διεθνών οργανισμών, αν δεν καταφέρουμε ουσιαστικά να προσαρμόσουμε τη δομή των οργανισμών προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε κίνητρα στους οργανισμούς για να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρούμε σε παράλληλες χρηματοδοτήσεις που ζητούν ουσιαστικά από τους πελάτες μας να συμπληρώσουν τα ίδια έντυπα χιλιάδες φορές. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις που θα μπορούσαν να δοθούν και που θα μας επέτρεπαν να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Σαφώς λοιπόν μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα στον τομέα αυτό και θα επανέλθω στο σημείο αυτό. Και τέλος, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουμε παρατηρήσει ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Η μεγάλη αυτή τράπεζα εξωτερικής χρηματοδότησης δανείζει, δάνεισε 9 δισεκατομμύρια ευρώ νομίζω πέρυσι. Είναι όσο μεγάλη είναι και άλλες τράπεζες διεθνής. Ορίμασε, αν θέλετε, η τράπεζα αυτή στα πλαίσια της παγκόσμιας τράπεζας, κινούμενη κυρίως ή υποκινούμενη μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υφίσταται λοιπόν πλέον, πατάει στα πόδια της, αλλά μεγάλωσε, ορίμασε με την οτροπία, αν θέλετε, της παλαιότερης τράπεζας στην οποία ανήκε. Δημιουργώντας λοιπόν μία νέα οντότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μία θηγατρική αν θέλετε, θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να γίνει κάτι τέτοιο, να δοθεί μία καλύτερη εξωτερική εικόνα στις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕΠ, έτσι ώστε η κουλτούρα της τράπεζας αυτή, η νοοτροπία της να τροποποιηθεί, να προσαρμοστεί καλύτερα, αν θέλετε, στις απαιτήσει των εξωτερικών δράσεων που καλείται να καλύψει. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα δίδει προς τους εταίρους τις πολύ καλύτερες υπηρεσίες, θα παρέχει πολύ καλύτερες υπηρεσίες, θα είναι σε άμεση επαφή με τους εταίρους αυτούς, θα μπορεί να αποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσει τους και επίσης εφόσον εγκρίνουμε τη νέα αυτή δομή, θα καταφέρουμε να, προσαρμοστούμε καλύτερα σε μελλοντικέ απαιτήσει, σε μια ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση της τράπεζας. Και έρχομαι κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Πρόεδρε, στις προοπτικές, τις μελλοντικές προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας μέχρι το 2020 όπου η εξωτερική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι όλο και πιο έντονη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όντω ναι, στα πλαίσια αυτού του νέου χρονοδιαγράμματος πρέπει να πάμε πιο μακριά και θα πρέπει να αναλύσουμε τις διαφορετικές επιλογές που έχουμε μπροστά μας προκειμένου να δώσουμε τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα αποτελεσματικό μέσο παρουσίας στο εξωτερικό, ισχυρής στεναρής παρουσία στο εξωτερικό. Δύο είναι οι βασικές επιλογές τις οποίες προτείνουμε αυτή τη στιγμή και οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν περισσότερο από τους ειδήμονες, οι οποίοι θα αποφαθούν τελικά πώς από νομικής και τεχνικής πλευράς μπορούν οι ε, προτάσεις αυτές να εφαρμοστούν. Πρώτον, θεωρούμε ότι οι αλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς να αυξηθούν η οικονομική πόρη χωρίς να αυξηθεί το κεφάλαιο το οποίο, θα, το οποίο εσείς θα πρέπει να δώσετε στις νέες δύο αυτές οντότητες που θα προκύψουν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι δύο αυτές οντότητες να λειτουργήσουν με ένα χαμηλό προπολογισμό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να φέρουμε μαζί καταρχάς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το τμήμα εκείνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων εξωτερικών δράσεων. Ουσιαστικά θα έχουμε αυτό το οποίο ονομάζεται στην ε, Παγκόσμια Τράπεζα LIDA, μια καλύτερη δηλαδή χρηματοδότηση, μια καλύτερη χορήγηση δανείων, μακροπρόθεσμων δανείων, που θα μπορούσε να γίνει με την καλύτερη συνεργασία των αρμοδίων τμήματων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι η ακόλουθη. Θα μπορούσαμε στο ίδιο πλαίσιο, στην ίδια δομή, να θέσουμε το σύνολο των ε, ταμείων εκείνων που συμβάλλουν στην εξωτερική χρηματοδότηση. Ο αναφέρομαι εδώ πέρα στο 63% του κεφαλαίου που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Λονδίνου, τη BERD. Θα βάζαμε επίση του πόρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εξωτερική Δράση. Θα θέταμε επίση στην διάθεση τη νέα αυτή δομή του πόρου τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώ επίση και του σχετικού πόρου του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Αν θέλετε, όλοι αυτοί οι χρηματοδοτικοί πόροι εξωτερική δράση, θα μπορούσαν να συγκεραστούν στα πλαίσια της ίδιας δομής. Θα είχαμε κατά αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη ορατότητα. Θα δημιουργούσαμε σίγουρα σε διεθνέ επίπεδο μια πολύ σημαντική μεγάλη δομή που θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί και στις νέες απαιτήσει που προκύπτουν από τη νέα διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε, όντως ήταν πολύ πλήρης η παρουσίασή σας και θα εξετάσουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με ιδιαίτερη προσοχή. Δίνω λοιπόν το λόγο τώρα στον εισηγητή μας, τον κύριο Κάλφιν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Καμντεσού για την έκθεση αυτή, καθώς επίσης και όλους τους συνεργάτες του από την Επιτροπή των Σοφών, από τη Στονιστική αυτή Επιτροπή. Η έκθεση αυτή δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα των στόχων που θα θέλαμε να πετύχουμε στα πλαίσια της εξωτερικής εντολής της Τράπεζα και γίνονται επίση και πολύ συγκεκριμένε προτάσει, οι οποίε νομίζω ότι θα προσελκύσουν πραγματικά το ενδιαφέρον μας. Αυτό είναι θέλετε το λιγότερο το οποίο μπορώ να πω σε αυτή τη φάση. Και όπω είπατε και εσεί, κύριε Καμπτεσιού θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε την νοοτροπία, τον τρόπο λειτουργία αν θέλετε τη Τράπεζα, όσον αφορά την εξωτερική τη εντολή, όσον αφορά τη χρηματοδότηση εξωτερικών δράσεων. Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτά τα οποία θα θέλαμε να πετύχουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσον αφορά την εξωτερική της εντολή, προκύπτουν πάντα κάποια ζητήματα, τα οποία συζητάμε συνεχώς. Καταρχάς, τα αποτελέσματα της εξωτερικής αυτής εντολής και πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δίδει προστιθέμενη αξία στα όσα γίνονται από άλλους φορείς, δηλαδή κυρίως σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική ανάπτυξη, με συγχωρείτε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το ζήτημα του προπολογισμού ανακύπτει συνεχώς. Αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε συνέργειες, δεν θα πρέπει να περιπλέκουμε ιδιαίτερα τα πράγματα, δεν θα πρέπει να δημιουργούμε παράλληλες δομές ή να χορηγούμε πόρους παράλληλα με χορήγηση ιδίων πόρων για συγκεκριμένες εξωτερικές δράσεις. Άλλα δύο ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά είναι το ζήτημα της διαφάνειας στην εργασία που κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συνεργάζεται με χώρες όπου το ζήτημα της χρηματοδότησης που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από άλλους ε, φορείς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Δηλαδή πρέπει να δίδει η χρηματοδότηση αυτή τα απαραίτητα αποτελέσματα. Πολλές φορές το διοικητικό περιβάλλον στις χώρες αυτές δεν είναι το ευκταίο και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνονται με πολύ προσεκτικό τρόπο αποφάσεις για το πόσα χρήματα ε, χορηγούνται και πώς ε, δαπανούνται τα χρήματα αυτά, πώς επενδύονται. Επίσης, κάθε φορά που μιλάμε για διαφάνεια θα πρέπει να μιλάμε και για ορατότητα. Και αυτό είναι ακόμα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δηλαδή, συνειδητοποιούν τελικά οι χώρες αυτές, στις οποίες πηγαίνουν τα χρήματα, ότι τα χρήματα αυτά αποτελούν τμήμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι χώρε αυτέ δεν είναι. ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι απλώ μια εμπορική τράπεζα που χορηγεί δάνεια, αλλά είναι μια τράπεζα που ουσιαστικά εξυπηρετεί την πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά λοιπόν που μιλάμε, και ιδίω τώρα που μιλάμε για την ενδιάμεση αναθεώρηση, θα πρέπει να έχουμε τα ζητήματα αυτά κατά νου. Ελπίζω λοιπόν να υποβληθούν σχετικέ προτάσει. Θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ περισσότερο σε κάποια από τα ζητήματα που άπτονται τη εξωτερική εντολή Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό φαίνεται ιδίω και στην έκθεση να υπάρχει ένα εσωτερικό συντονισμό στα πλαίσια δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τα διάφορα θεσμικά όργανα και Προτείνεται επίση να δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα όπου πολλοί ενδιαφερόμενοι εμπλεκόμενοι φορεί στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Ω προ την πρόταση αυτή, Εφόσον αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους ιδίου πόρους Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εφόσον πολλές φορές οι πόροι αυτοί έχουν να κάνουν με αποφάσεις που λαμβάνονται από διαφορετικές γενικές διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από αποφάσεις που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα κεντρικό συντονισμό. Πώς θα καταφέρουμε να διαρθρώσουμε το συντονισμό αυτό. ενδεχομένω ε, τα αποτελέσματα μερικέ φορέ να μην είναι απολύτω ικανοποιητικά. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες στην επιλογή των ε, κοινοτικών πόρων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και να μπορεί επίσης να συμβάλλει περισσότερο στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την χορήγηση χρηματοδότησης. Όσον αφορά τον εξωτερικό συντονισμό, συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών. Στη συνέχεια βέβαια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα μετά την πρόταση αυτή, γιατί ποιο αν θέλετε είναι ο επικεφαλής διεθνής χρηματοδοτικός οργανισμός στην περίπτωση αυτή, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα πώς θα εξασφαλίσουμε ότι ο ένας οργανισμός θα λάβει υπόψη του, ότι ένας οργανισμός θα λάβει του τους στόχους και τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η διεθνής αυτή συνεργασία πιστεύω ότι έχει και τους περιορισμούς της. Δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε να έχουν όλους τους στόχους, μάλλον όλοι οι διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί τους ίδιους στόχους και δεν θα καταφέρουμε να έχουμε τον ίδιο συντονισμό παντού. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε, κάποια κοινά πακέτα χρηματοδοτήσεων σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό, Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα. θα μπορούσαμε του οργανισμού αυτού να συνεργαστούμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουμε κοινού στόχου σε πολλού τομεί, μικρομεσαίε επιχειρήσει, υποδομέ, κλιματικέ αλλαγέ ε, κτλ. Ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στου τομεί αυτού να είχε πιο ηγετικό ρόλο. Πάντω νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν κάποια κοινά πακέτα εντό αγωγικών χρηματοδότηση όπου θα μπορούσε η ΕΤΕΠ να συνεργάζεται με άλλου διεθνεί χρηματοδοτικού οργανισμού. About... Όταν μιλάμε για αποτελέσματα τώρα. Καλό είναι να ρωτάει κανεί, εντάξει είναι αρκετά ικανοποιητικό, μα ικανοποιεί το τι κάνει η τράπεζα. Πρώτο όμω πρέπει να δούμε την κατάσταση εκτενέστερα. Είναι ικανοποιητικά τα κονδύλια που ξοδεύονται από το προπολογισμό τη Ένωση. Αν ζητάμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει επίση να δούμε και πώ ε, χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκοί πόροι ανάπτυξη στι ίδιε χώρε και μετά να δούμε τι συνέργειε και να πούμε τι είναι αποτελεσματικό, τι δεν είναι, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι είμαστε κάπως πιο επικριτικοί στον τρόπο χρησιμοποίησης των, του Ταμείου Ανάπτυξης από την Ένωση. Και ίσως θα έπρεπε να δούμε το ενδεχόμενο να διευρύνουμε το σύστημα. Κάτι άλλο. Το αναφέρατε στην έκθεσή σας οι στόχοι. πάνω στους οποίους δουλεύει η ΕΤΕΠ στην, στο εξω, στις εξωτερικές δραστηριότητες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιβάλλον, ανάπτυξη. Αλλά η ανάπτυξη διάφορες χώρες και το γεγονό ότι ε, και οι συνέπειες που θα έχουν οι επενδύσεις ή οι δωρεές αυτές με οδηγούν στην εξής ερώτηση. Μπορεί η τράπεζα να έχει έναν πιο ε, δραστήριο ρόλο στην εκπαίδευση, στην υγεία. Ξέρουμε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα κάνει μια καλή δουλειά στον τομέα αυτό. Και αυτό δεν είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνουν άλλοι ε, αναπτυξιακοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Στην έκθεση αναφέρεται ότι μπορεί να το εξετάσετε στην ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά να δείτε και πώς τα προγράμματα επηρεάζουν την εκπαίδευση εκπαίδευση, την καταπολέμηση της φτώχειας σε καθημερινότητα της, των χωρών. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε τέτοιες ε, συνέργειε όταν μετρούμε τον αντίκτυπο των, Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Εντέψης στις χώρες αυτές. ακόμα, μερικές ακόμα παρατηρήσεις. Σίγουρα θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και άλλη φορά. Είναι κρίσιμο να βρούμε τρόπο για να εμπλακούν και άλλοι φορεί, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνεί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, αλλά και οργανισμοί του συστήματος του ΟΗΕ, η UNICEF για παράδειγμα, που έχουν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, η Ερυθρά Έλληνος, που έχουν προγράμματα συναφή στις χώρες εκείνες αλλά να ανοιχτούμε και σε κάποιους μικιό, που μερικές φορές είναι αρκετά επικριτικές εναντί της ΕΤΕΠ. Αναγνωρίζοντα ωστόσο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια στη δουλειά τη τράπεζα. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ε, εντονότερα, δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων στις ε, συζητήσεις. Ένα από τα θέματα που πρέπει να αποφασίσουμε είναι η εντολή για τα δύο δις. Είπε ο κύριος Καμπντεσίου ότι έχουν ε, διοχειρευτεί τα κονδύλια χρησιμοποιούνται για περιβαλλοντικά θέματα, δεν σχετίζονται με τα ανώτατα όρια που υπάρχουν. Η πρόταση είναι ενδιαφέρουσα, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε. Αρκεί το περιβάλλον. Αρκεί να πούμε ότι διασπείρουμε τα κονδύλια παντού. Γιατί 2 δισεκατομμύρια δεν είναι πολύ σημαντικά για να πετύχεις ε, ένα συγκεκριμένο στόχο. Να δούμε και την περιφερειακή διάσταση, πώς κατανέμονται περιφερειακά και την ουσία. Πώς χρησιμοποιούνται στην πράξη. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω στην έκθεση Σωστά αναφέρεται ότι στις χώρες αυτές η διοικητική ικανότητα είναι αδύναμη και προφανώς μια δουλειά είναι η ενίσχυση της ΕΤΕΠ, είναι η ενίσχυση της διοικητικής υποδομής, αλλά μήπως εδώ θα έπρεπε να εξετάσουμε και το δεχόμενο καλύτερο συντονισμό με, τις, ε, με την εξωτερική διπλωματική υπηρεσία της Ένωσης, τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορούν να δώσουν Συμβουλή. Δεν είμαι βέβαιο ότι η ΕΤΕΠ θα μπορεί να θεσπίσει, να έχει μια πολύ στενή παρακολούθηση του τι γίνεται στις ε, ε, δικαιούχου χώρε, όσο και να αυξήσει κανεί το προσωπικό του, το προσωπικό της Τράπεζα. Εντάξει, αύξηση του προσωπικού, αλλά α δούμε και πώ άλλες συνέργειε στην Ένωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Τελειώνω, Πρόεδρε. Γιατί ξέρετε ότι έχετε πολλή δουλειά και δύσκολη δουλειά προσπαθώντας να κρατήσετε το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε πολλά θέματα που συζήτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Καμπτεσού για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στον τομέα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Νομίζω ότι η εισήγηση του κύριου Καμπτεσού επέτρεψε να ξεκινήσει μια καρποφόρα συζήτηση που και εσείς το φορτήσετε σε λίγα λεπτά θα σταματήσουμε δυστυχώ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο εισηγητή αντιπρόεδρο κ. Καλφίν, θέλω να επιστήσω την προσοχή σε ένα θέμα που μέχρι τώρα δεν είδαμε παρκώ, ούτε καν εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών. Τον συντονισμό μεταξύ των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των διεθνών ε, δανειστών. Ένα εξίσου σημαντικό θέμα υπάρχει που δεν το είδαμε. Το συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών, διότι ο προπολογισμό της Ένωσης, ο 9, 8 με 9 δις προπολογισμό της Ένωσης και ΦΕΔ είναι, πηγαίνουν στην αναπτυξιακή βοήθεια. Αν όμως αφήσουμε και τους εθνικούς προπολογισμού των 27 χωρών για την ανάπτυξη, φτάνουμε σε δεκαπλάσια ποσά. Ο συντονισμό μεταξύ των προσπαθειών αυτών, των 28 αυτό προπολογισμών στην πραγματικότητα, γίνεται θεωρητικά στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Ανάπτυξης, αλλά επιτόπου, πολύ άσχημα υλοποιείται. Και σίγουρα ένα από τα βασικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, παράδειγμα είναι η πολιτική ανάπτυξη, υπάρχουν και άλλοι παρόμοιοι τομεί, τελείω διαφορετική έρευνα π.χ. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσουμε όταν μελετούμε την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προ προοπτικών για την χρηματοδότηση των κοινών ευρωπαϊκών στόχων τα επόμενα έτη, θα είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε καλύτερα ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί συνδράμουν επίσης τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κοινών στόχων. Κάθε φορά λοιπόν που εθνικός προϋπολογισμός εφαρμόζεται σε κοινό στόχο, να εξασφαλίζουμε αυτόματα ότι θα υπάρχει μια συνέργεια, μια, ένα συντονισμός και όχι μια διασπαρμένη ή και αντιφατική δράση. Να υπάρχει λοιπόν ένα blending μεταξύ δανείων και ενισχύσεων, μεταξύ διαφορετικών τεχνικά μορφών χρηματοδότησης, αλλά και ένα Εξίσου σημαντικό, εξίσου σημαντικό είναι το πολιτικό blending. Θέλει κάποια σχόλια να κάνει ακόμα ο κύριος Καμπτεσί και ίσως να κλείσει και ο κύριος Μιστάτ. Μισελ. Εκτός μικροφώνου. Για το τελευταίο θέμα, Πρόεδρε, μεταξύ των προτάσεών μας, ήθελα να το πω αλλά δεν πρόλαβα, προτείνουμε να υπάρξει μια πλατφόρμα στην οποία θα γινόταν αυτό το blending όχι μόνο από την Επιτροπή και την ΕΤΕΠ αλλά και διμερείς δωρητές οι μεγάλες χώρες, ούτως ώστε να υπάρξει ακόμα καλύτερο συντονισμός και ακόμα μεγαλύτερη συνέργεια. Δύο-τρία πράγματα να πω για τα δύο δις. Όντως πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να στραφούν προς ε, την αλλαγή του κλίματος. Η περιφερειακή κατανομή θα πρέπει να γίνεται με βάση τα σχέδια που υποβάλλονται, αλλά τα δύο δις θα δώσουν κάτι αρκετά σημαντικότερο, γιατί αν προσθέσουμε και άλλα τρία που θα δώσει η ΕΤΕΠ ως δάνειο από τους δικούς της πόρους, φτάνουμε στα 5 και σε αυτό θα προσθεθούν τα 7 δις σε ετήσια βάση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αλλά μιλάμε για τρία πακέτα μαζί που οδηγούν σε πολύ πιο αξιόπιστες δράσεις και προφανώς η ικανότητα ενισχύσεων από την Επιτροπή θα επιτρέψει όχι μόνο ε, δραστηριότητες μετριασμού αλλά και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος στις φτωχές χώρες σε συνέργεια με το πακέτο ανάπτυξη. Μια τελευταία παρατήρηση. Και δεν θέλω να σας κολακεύσω. Μεταξύ των μεγάλων αλλαγών της τελευταίας δεκαετίας περιλαμβάνεται και ο ρόλος του Κοινοβουλίου η ομάδα μας διαπίστωσε ότι δύο τομείς στους οποίους είναι αποφασιστική η παρέμβαση του, κοινο, του Κοινοβουλίου ήταν η συνένεση για την ανάπτυξη. Εδώ ξεκινάει και η πολιτισμική προσαρμογή της τράπεζας, η προσαρμογή της ένα δηλαδή περιβάλλον σε ένα χώρο που δεν την ενδιαφέρει κατά προτεραιότητα μέχρι τώρα. Επίσης να σας πω ότι το ότι τονίσαμε να κάνουμε προτάσεις για το μέλλον, μια ιδέα για μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Ε, ε, το κάναμε γιατί η έκθεση Μίτσελ πριν από δύο χρόνια μας παρότρινε να σκεφτούμε για να φέρουμε πιο κοντά και πιο οργανικά κοντά την ΕΤΕΠ και την ΜΠΕΡΤ Εδώ σταματάω. Ο κύριος Πέρμαν ήθελε να μιλήσει για 30 δευτερόλεπτα. Ήμουν δημοσιογράφος 20 χρόνια. Μπορώ να μιλήσω λοιπόν 2 λεπτά, αλλά 30 δευτερόλεπτα είναι λίγο. Ως εισηγητής για την εξωτερική εντολή της ΕΤΕΠ από την Επιτροπή Ανάπτυξης θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είναι πολύ σημαντική και εξαιρετικά επίκαιρη η έκθεσή σας εν μέση οδό της αναθεώρησης της εντολής ε, που θα μας επιτρέψει να συμπεριλάβουμε πολλές από τις συστάσεις σας στην έκθεσή μας. Προφανώς υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση. Λέτε ότι πρέπει να γίνει μια πραγματική τράπεζα ανάπτυξης αυτό που ζητάτε στην πραγματικότητα. Αλλά εδώ έρχεται σε ανταγωνισμό με την Παγκόσμια Τράπεζα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με 26%. Άρα μήπως μια συζήτηση που θα μπορούσε, θα μπορούσε να είναι τι θέλουμε καλύτερα. Θέλουμε να ενισχύσουμε την Παγκόσμια Τράπεζα ή θέλουμε μια δική μας Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Εγώ είμαι ε, Ευρωπαίος ε, με πεποίθηση. Πιστεύω ότι ε, πρέπει να έχουμε ένα δικό μας εργαλείο, αλλά μήπως τελικά φτάσουμε σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των δύο στόχων που επιδιώκουν τους ίδιους στόχους. Μείωση τη φτώχεια. ένταξη όλων των πολιτών του κόσμου, οικονομική ένταξη, πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στα δάνεια, στην αποταμίευση, στην ασφάλιση. Αυτά τα τρία πράγματα είναι καθοριστικά. Ήμουν σε μια συνάντηση με βοσκούς από το Σαχέλ και μου έδωσαν αυτό. Δεν, μην με ρωτήσετε τι είναι. Ε, είναι. Από ε, χαλκό. Για να γίνει αυτό χρειάζεται όμως λεφτά. Χρειάζονται ε, μια σειρά υποδομών. Κατόπιν, δύο πράγματα. Η ΕΤΕΠ είναι τρομερά δειλή. Μιλάτε για διαφορετικές αλλαγές, αλλά αυτές οι αλλαγές τις βλέπετε από πάνω. Η βοσκή αυτή θέλουν πρόσβαση και η πρόσβαση γίνεται από κάτω. Αυτό είναι που λείπει από την έκθεση και αυτό είναι που λείπει και από την ΕΤΕΠ που ασχολείται με τους μεγάλους εμπλεκόμενους, όχι με τους πολίτες. Άλλο η Ευρώπη. Στην Ευρώπη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η ΕΤΕΠ είναι αναγκαία. Μπορεί να μην το ξέρουν αλλά είναι αναγκαία. Αλλά έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε για, τους, αν, για τις αναπτυσσόμενες χώρες και είμαι πεπισμένος ότι η ΕΤΕΠ μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και σε τραπεζικές υποδομές και σε δικτύωση τοπικών τραπεζών με υποστήριξη της ΕΤΕΠ που προφανώς δεν πρέπει να δημιουργήσει δικούς της εκπροσώπους και όλα αυτά με σεβασμό των στόχων που αναφέρεται. αλλαγή κλίματος, βιώσιμη οικονομία, τοπική κουλτούρα, κάτι που το απαιτεί άλλωστε και η συνθήκη της Λισαβόνας. Η ειδηλή αυτή της ε, ΕΤΕΠ εμφανίζεται κυρίως όταν μιλάμε για μικροχρηματοδότηση. Από τα 10 δις, μόνο 90 εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί σε μικροδάνεια. Πολύ λίγο. Και πιστεύω ότι οι υπάλληλοι της ΕΤΕΠ θα ήθελαν να το αλλάξουν αυτό. Εμείς όμως πρέπει να τους το ε, επιτρέψουμε. Όχι ντε και καλά να πάμε στον κάθε κάτοικο του Μαλή, αλλά να χρησιμοποιούμε τη να προσφέρουμε τη δυνατότητα ε, σε τοπικές τράπεζες, σε ομάδες πολιτών που έχουν τη δυνατότητα, που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβαση σε άλλη τράπεζα, να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Μεσάντα μπορεί να ολοκληρώσει, αλλά θα ήθελα να πω ότι προφανώς όταν έχουμε επικαλύψεις, όπως είπατε και εσείς, το θέμα είναι οι Ευρωπαίοι χρηματοδοτούν τη διαφορά. Και από την Διεθνή Τράπεζα οι Αμερικανοί ωφελούνται πολιτικά. Εάν οι Ευρωπαίοι εφαρμόζοντας αυτό που θα έπρεπε να έχουν κάνει από τότε που έχουμε τη συνθήκη της Μαστρίχ, με την ενθάρρυνση της συνθήκης της αγώνας και υπό την αιγίδα του πρόεδρου Φανρόπεϊ αποφάσισαν να μιλήσουν με μία φωνή σε όλα τα βήματα διεθνών οικονομικών διαπραγματεύσεων θα υπήρχαν σημαντικές οικονομικές αλλαγές και οι απλουστεύσεις θα ε, δημιουργούνται από μόνοι Ο πρόεδρος κ. Μέσσατ έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίε να συζητήσουμε τα ίδια θέματα. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όλες οι στάσεις τη επιτροπή που αφού αποφασίζονται για βραχυπρόθεσμο τομέα, με μία εξαίρεση, είναι καλό. Η μόνη εξαίρεση είναι τα επιχειρήματα που λένε θα πρέπει να έχουμε μία θηγατρική. Καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία του κ. Καμπιουσί που πιστεύει ότι θα μπορέσει να γίνει αυτή η σημαντική αλλαγή συνηθιών, ότι όταν παρεμβαίνουμε δηλαδή στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την ίδια τακτική που έχουμε στο εσωτερικό της ε, Ένωσης, καταλαβαίνω γιατί αυτό μπορεί να είναι σωστό, αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα. Όλες οι άλλες συστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες, είναι καλόδεκτες ίδιος η σύσταση να απλουστεύσουμε και να αναγνωρίσουμε τους όρους εξωτερικής αίτηση, γιατί είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε σε κάποιον, στον ίδιο, ότι μπορούμε αυτό να το κάνουμε στη μία περιοχή και να μην το κάνουμε στην άλλη, γιατί αυτό το μέσο μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε σε μία περιοχή και στην διπλανή. Λοιπόν, να εναρμονιστούν οι εντολές. Αυτό θα ήταν θαυμάσιο. Το ίδιο και η σύσταση να έχουμε κάθε χρόνο λειτουργικές οδηγίες που ορίζονται με συμφωνία μεταξύ της Κομισιόν και της ΕΤΕΠ. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ρεαλιστική ε, προσέγγιση για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ευθυγράμμιση και την συνοχή και των μέσων και των στόχων. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η σύσταση τα δύο δις που ήταν στο αποθεματικό να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλογών, μου φαίνεται απόλυτα δικαιολογημένο. Πραγματικά επιβεβαιώνω ότι οι βραχυπρόθεσμε συστάσεις είναι όχι μόνο αποδεκτέ, αλλά και καλότακτες από την ΕΤΕΠ. Τώρα το δεύτερο τμήμα τη έκθεσης που αφορά τι πιο μακροπρόθεσμες ε, συστάσει. Δεν θα το αναπτύξω ιδιαίτερα σήμερα, αλλά θέλω να σα πω ότι αυτό το δεύτερο τμήμα γύρει σημαντικά θέματα, πολύπλοκα θέματα και οι πρώτε αντιδράσει οι δικέ σα, κύριε Πρόεδρε και εκείνες του κύριου Μπέρμαν, καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η θα υπάρχει πραγματικά συζήτηση. Συζήτηση που ελπίζουμε να είναι εις βάθος. Αυτή τη στιγμή, όχι σαν άποψη της ε, ΕΤΕΠ, αλλά σαν Ευρωπαίος πολίτης, θα είχα να πω ότι συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες στις οποίες βασίζονται οι συστάσεις της Επιτροπής Και Την ανησυχία δηλαδή να ενδυναμωθεί η συνοχή, η αποτελεσματικότητα και η οραματικότητα της ε, δράσεις της ΕΤΕΠ. Αν το συζητούσαμε δύο μακρόν θα μπορούσα να σας δώσω πολλά παραδείγματα όπου χάνουμε αποτελεσματικότητα και πολιτική οραματικότητα λόγω της έλλειψης συντονισμού, λόγω του ότι ο καθένας Ευρωπαίος ε, ε, παράγοντας δρά διαφορετικά. Υπάρχει λοιπόν ένα κοινό ενδιαφέρον να ενδυναμώσουμε την συνοχή, την αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι κάτι που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Η Επιτροπή έκανε κάποιες συστάσεις, αρκετά ριζοσπαστικές, αλλά πιστεύω ότι θα είναι καλό να τις εξετάσουμε εις βάθος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα, σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Πρόεδρε. Γεια, ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ορατές οι δράσεις της ΕΤΕΠ. Άκουσα κάποιον Γάλλο να λέει κάποια στιγμή. Ε, ένας άνθρωπος πολύ ικανός είπε για το πρόεδρο μας, αλλά έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα πολιτικά. Είναι μετριοπαθής. Ο κύριος Μάισατ είπε ότι είναι πάρα πολύ μετριοπαθής, είπαμε. Ε, λοιπόν, θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να είναι καλύτερα γνωστή η ΕΤΕΠ, η οργάνωσή της, ε, η λειτουργία της και οι συστάσεις της. και είναι σίγουρο ότι αυτά που προτείνει η Επιτροπή Καντούση θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι μια πρώτη ενταλλαγή απόψεων. Από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει βέβαια να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, να υποβάλει κάποια σύσταση και βάσει αυτή θα μπορέσουμε επίσημα να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε αυτόν τον διάλογο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προσθέσετε απόψε στην πρώτη αυτή ενταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Merci. Voilà. Karl Bien, alors, euh, les vice-présidents qui étaient restés modestement bas. Λοιπόν, οι, πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι που είχαν μείνει εκεί με τρεπαθώς μπορούν να περάσουν στο έδρανο για να είναι και πιο ορατοί. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης. 5 και 6 μάλιστα. Μια ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες ε, της ε, προβλησμού της Επιτροπής για το 2011 με ένα έγγραφο εργασία που είχαμε μια πρώτη παρουσίαση από τη Συνδονία για Ντέτσκευσκα και μετά το σχέδιο έκθεση. Συντονία, έχετε το λόγο. Ε, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, E, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας παρουσιάσω τις ε, ε, δημοσιονομικές προτεραιότητες. Όπως δικαίως είπατε, Υπάρχει ένα θέμα που ήδη συζητήσαμε στην περασμένη συνεδρία της ε, Επιτροπής Προπολογισμών. Ήδη δηλαδή αναφερθήκαμε στο έγγραφο εργασία που αναφέρεται στην εισαγωγή της συνθήκης Αβώνα, στην ετήσια δημοσιονομική διαδικασία. Εγώ θα περιοριστώ λοιπόν στην παρουσίαση των νέων στοιχείων. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα περιοριστώ σε δύο σημαντικά μηνύματα που περιλαμβάνει αυτό το έγγραφο. Γιατί πρόκειται για ένα πολύ αναλυτικό έγγραφο και γι' αυτό θα προσπαθήσω να περιορίσω τις προτεραιότητες σε λίγες μόνο, σε λίγα σημεία. Ήταν δύσκολο όμως να αντισταθώ στον πειρασμό και στην επιθυμία των συναδέλφων να υπάρχουν περισσότερες από αυτές τις προτεραιότητες. Θα θυμόσαστε ότι είχα πει κάποια στιγμή ότι θέλω να περιοριστώσω τις προτεραιότητες αυτές όπως λέει από αυτής θα, θα θείτε απογοητευμένοι γιατί έχω διευρύνει το έγγραφο. Η διεύρυνση αυτή ήταν όμως τυχαία. Ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησής μου στο Στρασβούργο με τις δικαιωμένες ε, επιτροπές και τους ε, διάφορους ε, υπεύθυνους για θέματα δημοσιονομικά και τους εισηγητές που μου έδωσαν κάποιες ιδέες που, ανάσκα, που αισθάνθηκα ότι πρέπει αναγκαστικά να συμπεριληφθούν. Θα ήθελα να σας απτύξω δύο κυρία θέματα. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω ότι οι πολιετής προοπτικές που είχαν υιοθετηθεί το 2006 τώρα φτάνουν στα όρια τους. Τα περιθώρια ελισμού που έχουμε εξ αυτού είναι πάρα πολύ μικρά. Αυτό το αναπτύσσω για άλλη μια φορά στην πρότασή μου για τις δημοσιογικές προτεραιότητες. Και δυστυχώς ε, αυτή είναι μια λυπηρή πραγματικότητα που θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου. Οι πολιτικές προοπτικές έχουν ήδη ανα... επανεξεταστεί τέσσερις φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε αυτό και το επόμενο έτος θα έχουμε έλλειψη πόρων. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ένα από τα όνειρά μου για το 2011. Θα ήθελα να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της νεότητας, νεότητας με την ευρύτατη έννοια. Δηλαδή κυρίως στην χρονική στιγμή κάθε ε, ε, ανθρώπου κατά την ε, χρονική στιγμή της ζωής του, την οποία μεταβαίνει από την εκπαίδευση στον χώρο εργασίας. Η νεότητα είναι κάτι που συνδέεται συνήθως με τη μάθηση, με την παιδεία. Εγώ θα ήθελα να εξετάσω τι προβλέπει ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή για του νέου και τι θα μπορέσουμε να διορθώσουμε και να προσθέσουμε, να του προτείνουμε περισσότερα πράγματα τμήμα λοιπόν της κοινής μας εργασίας ε, θα είναι να εξετάσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένα προγράμματα πιλότους που αφορούν κυρίως τους νέους. Όπως είπα ήδη, στις επαφές που είχαμε στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές συνέλεξα συμπληρωματικά στοιχεία για το έγγραφό μου αυτό το έγγραφο εξακολουθεί να είναι ανοιχτό. Δεν ήθελα να σας υπενθυμίσω το τι πρέπει ακόμα να κάνουμε. Μέχρι τις 25 τρέχοντας μπορούν να υποβληθούν ε, τροπολογίες για τις ε, προτεραιότητες. Περιμένω λοιπόν να ενισχύει να ακούσω τις ε, προτάσεις σας και τις ιδέες σας. Γιατί έχω ακούσει τις ιδέες σας, αλλά όχι όλων τις ιδέες. Περιμένω να ακούσω και τις ιδέες των άλλων για να μπορέσω να τροποποιήσω το έγγραφό μου και ελπίζω να υιοθετηθεί στην Ολομέλεια, τη δεύτερη Ολομέλεια του Μαΐου. Επίσης θα επιθυμούσα το έγγραφο αυτό να θεωρηθεί σαν ένα πρώτο κείμενο για το έτος 2011. Γιατί μια που έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να μας υποβάλει τις ε, δημοσιομικές της προτεραιότητες. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε από κοινού να προετοιμάσουμε εδώ την άποψη του Κοινοβουλίου και να την υποβάλουμε κατά όπως μοναστικό τρόπο το φθινόπωρο όταν θα έχουμε το κοινό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να το έχουμε κατά νου όταν συζητάμε τα θέματα αυτά. Δηλαδή, ο προπολογισμό του 2011 είναι ένας πάρα πολύ ιδιάζων προπολογισμό, γιατί πρόκειται για τον πρώτο προπολογισμό που ακολουθεί τις συστάσεις της συνθήκης τη και είναι μια πρώτη δοκιμή για να δούμε κατά πόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δεύτερον, θεωρούμε ότι θα πρόκειται για μια τελική δοκιμή πριν αποφασίσουμε για τις δημοσιονομικές προβλέψεις για μετά το 2013. Γι' αυτό είμαι πεπισμένη ότι το προϋπολογισμό του 2011 είναι πολύ ιδιάζον και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και βασίζομαι στις προτάσεις σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ Συντονία. Δικαίως αναφερθήκατε στην πολιτική σημασία αυτού του προπολογισμού. Και αισθανόμαστε πραγματικά ιδιαίτερα ευτυχεί που ένα τόσο ικανό άνθρωπο όσο εσεί έχει αναλάβει τον προπολογισμό αυτό. Γιάννη Γιάννη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ Σιδονιά για μια πάρα πολύ καλή εργασία και για το έγγραφο εργασία το οποίο θα θέλω να αναφερθώ αυτή τη στιγμή. Το έγγραφο εργασία για τη διαδικασία αντικατοπτρίζει και το γεγονό ότι έχουμε τη νέε διαδικασίε συνθήκη Λισαβόνα, αλλά και ότι εσωτερικά είχαμε κάποιε μεταρρυθμίσει. Πολλοί από εμά που ήταν παρόντες όταν έγινε αυτό ο ιδιαίτερα, θα θυμόσαστε πόσο δύσκολο ήταν πολλές φορές να εξηγήσουμε σε άλλους βουλευτές τι σημαίνει η δημοσιονομική αυτή διαδικασία. Και ότι καμιά φορά είναι διαφορετική από τις νομοθετικές διαδικασίες. Θα ήθελα να φέρω ένα τεχνικό θέμα που είναι όμως τεράστια σημασία νομίζω για όλες τις πολιτικές ομάδες. Στη σελίδα 4 ή 5, ανάλογα με τη γλώσσα που θα παρακολουθήσετε, υπάρχει το θέμα της διαδικασία ε, διαδικασίας συνδιαλλαγής και είχαμε πολλές συζητήσεις για το πώς θα πρέπει να γίνει αυτό γιατί υπήρχε μια τάση στο κοινοβούλιο να λέγεται ότι θα πρέπει να ακολουθήσει τη συνήθεια διαδικασία διαλλαγή. Ενώ αυτό ήταν πάντα αρμοδιότητα τη Επιτροπής Προπολογισμών και χρησιμοποιούσαμε ακριβώς όλο το έτος για να προετοιμαστούμε για αυτή τη συνδιαλλαγή. Να επαναλάβουμε τα επιχειρήματά μας, να ξέρουμε τους κανόνε, κλπ. Θα λοιπόν να είμαι σίγουρη ότι η διατύπωση αυτή σημαίνει ότι εξακολουθούμε να είμαστε στην κατάσταση στην οποία εμείς αποφασίζουμε για τη διαδικασία, ενώ βέβαια ο πρόεδρος μαζί με τον εισηγητή είναι εκείνος ο οποίος ε, λαμβάνει μέρος στις διαπραγματεύσεις. Το αγγλικό κείμενο είναι κάπως διαφορετικό από τα άλλα που λέγεται. Μια μικρή ομάδα προετοιμάζει την απόφαση. Θα έπρεπε να είναι μάλλον ότι προετοιμάζει την πρόταση για την απόφαση. Έχουμε μια μικρή ομάδα με τον πρόεδρο, στον εισηγητή και στο συνειδητικό ειδικό ε, εισηγητή γιατί καμιά φορά χρειάζεται κανένας να επισέλθει στις λεπτομέρειες. Είναι καλό, παραδείγματος χάρη, να έχουμε κάποιον που γνωρίζει το θέμα σε όλες τις λεπτομέρειες και όταν έχουμε συναπόφαση εδώ θα πρέπει εκείνοι που έχουν βοηθήσει στην λήψη της, απο... της ε, απόφασης για την πρόταση να είναι παρόντες. Γιατί εμείς είμαστε βουλευτές, γιατί είμαστε πιο ευφύς από το Συμβούλιο και θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να είναι σίγουρο ότι η ερμηνεία αυτών που λέγονται εδώ να ακολουθεί αυτό που είδαμε να λαμβάνει η χώρα τα περασμένα έτη και να υπάρχει έτσι μια, ένα ανοιχτό πνεύμα στις αποφάσεις που επιδιώκαμε πάντα. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Πολύ ξεκάθαρα αυτά. Η Γιούτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την τελευταία παρατήρηση τη Άννη, δεν θέλω να προσθέσω πάρα πολλά, γιατί ξέρω ότι το συζητήσαμε αυτό και στην ε, ε, ομάδα εργασία τη ομάδα μου και υπάρχουν ορισμένοι που έχουν κάποιες ιδέες για το τι θα μπορέσουμε να έχουμε εδώ κατά νου. Και πρόκειται και για το θέμα της εντολής που θα πρέπει να έχει αυτή η ομάδα εργασία. Κατά πόσο είναι είτε 20 είναι 20 ή 3 είναι το ίδιο. Θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη εντολή. Εγώ θα ήθελα να πω στη Ζητωνία ότι το έγγραφο για τις προτεραιότητες το έκανε καταπληκτικά. Και εγώ το ξέρει και αυτοί που με ξέρουν Είμαι πάρα πολύ φιδωλή με, επεν, με επένους, αλλά θα πρέπει να πω πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ καλό το έγγραφο αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, συμφωνώ ότι θα πρέπει πραγματικά, όπως λέγεται στον τίτλο, να περιορίσουμε, να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις προτεραιότητες. Ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι θεωρούν πολλά πράγματα σημαντικά και για τον προπολογισμό 2011. Είναι και πολλά πράγματα σημαντικά. Δεν το συστάμε, αλλά θα πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά και στη συνδιαλλαγή. Είτε τα εγγράψουμε τώρα εδώ στις προτεραιότητες, είτε όχι. Γι' αυτό, εάν διατυπώσουμε πιο προσεκτικά το τι εννοούμε με το θέμα αυτός της πολιτικής για τους νέους, θα ήταν καλό να το ανεπτύξουμε λίγο παραπάνω από αυτό που ε, λέει η Σιδονία. Τώρα, εγώ επέμεινα να λέμε προτεραιότητες, προτεραιότητες και να μην αλλάξουμε τίποτα, αλλά όμως κάτι θέλω να πω. Θέλω να υπάρχει μια παράγραφος για τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης των κλιματολογικών αλλαγών. Ακριβώς μετά από αυτά που ακούσαμε από την ΕΤΕΠ μόλις τώρα, αυτά που είπε ο κ. θα πρέπει κάπου να υπάρχει μια παράγραφος που να λέει και αυτό θα πρέπει τώρα να ξεκινήσει. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε πρέπει το 2011. Γιατί αυτό δεν θα είναι μια προτεραιότητα μόνο για το 2011, αλλά για το μέλλον οπωσδήποτε. Αν οπωσδήποτε κάτι πρέπει να κάνουμε. Κατά τα άλλα έχω πάρα πάρα πολύ μικρές ε, παρατηρήσεις, θα σας στείλω. Καμιά φορά μια λέξη ίσως ή κάποια διευκρίνηση. Άμα μιλάς για την εξωτερική ε, υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων, θα πρέπει να πούμε ότι βέβαια χρειάζονται πόρους, αλλά διοικητικούς πόρους, για να είναι σαφές τι έχουμε κατά νου. Πώς θα πρέπει να προηγουμένει αυτή η υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων. Ότι δεν πρέπει δηλαδή να έχουν λειτουργικούς πόρους για να κάνουν και δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η απόψή μου τέλο πάντων. Και ελπίζω ότι και εδώ όταν το συζητήσουμε το θέμα θα μπορέσουμε να βρούμε τη λύση. Κατά τα άλλα το βρίσκω πραγματικά θαυμάσια ότι δεν πρόκειται για απλές κατηγορίες γραμμές αλλά για προτεραιότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci, Σε ευχαριστούμε, Γιούτα. Όντω η Γιούτα έχει δίκιο και κάνει πολύ καλά που αναφέρεται στην χρηματοδότηση της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Για να μην επιμικίνουμε πάρα πολύ τη συζήτηση, δεν απάντησα στα όσα είπε ο κύριος Καμπτεσιού, όταν αναφέρθηκε όμως τα δύο αυτά δισεκατομμύρια τα οποία θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δώσει στην πολιτική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, είχε πει ότι θα έρθουν επιπλέον στα 3,7 δισεκατομμύρια τα οποία θα δώσει ο κοινοτικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα την πρόταση αυτή και από ευγένεια δεν τον διέκοψα βέβαια. Δεν του είπα ότι εμεί ουσιαστικά θα αποφασίσουμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Όντω όμω από την Κοπενχάγη τα πράγματα τα συμπεράσματα ήταν αρκετά σαφή. Θα δούμε τι θα προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να δούμε το ζήτημα αυτό και να δούμε τελικά ποιες πολιτικές επιλογές θα γίνουν για τον προπολογισμό του 2011. Προτείνω για την Επιτροπή, η Επιτροπή Προπολογισμό να γίνει για μια στιγμή η Επιτροπή Γυναικών στη συζήτηση της έκθεση στη συντονία, γιατί μόνο γυναίκες νομίζω θέλουν να πάρουν το λόγο. Μετά τη Γιούτα λοιπόν, η κυρία Μπαλτσάνη θέλει το λόγο και τη τον δίνω αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Οι επιλογές της Συντόνια με βρίσκουν σύμφωνοι. Δηλαδή, το ότι θέλουμε να έχουμε ένα σημαντικό ποσό, ένα σημαντικό κονδύλιο για την πολιτική νεολαία του 2011. Και θα μπορούσε το ζήτημα αυτό να συνδεθεί και με άλλα σημαντικά ζητήματα όπως η κινητικότητα, επιχειρηματικότητα, η κατάρτιση και η εκπαίδευση. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να υπογραμμίσουμε για ποιο λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να θέσει την πολιτική για την νεολαία σε πρώτη θέση. Νομίζω θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε δύο βασικές κατευθύνσεις. Πρώτον, πολιτικές υποστήριξης των νέων, οι οποίες βρίσκονται στη βάση οποιασδήποτε κοινωνικής πολιτικής που έχει ως στόχο την ένταξη, την ενσωμάτωση των ε, πολιτών. Αν θέλει πραγματικά να προωθήσει κανείς την ανεξαρτησία, την ε, δυνατότητα των ανθρώπων να εργάζονται, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι μας είναι ενσωματωμένοι και ότι τους υποστηρίζουμε δεόντως. Και για ένα όμως λόγο πρέπει να υποστηρίξουμε τους νέους είναι αυτοί που έχουν τον τεράστιο αυτό ταλέντο της ε, καινοτομίας. Αν δημιουργήσουμε λοιπόν τις κατάλληλες συνθήκες, οι νέοι μπορούν να αποτελέσουν μια πραγματική κινητήρια δύναμη. Μιλάμε συνεχώς για την πράσινη οικονομία. Για ποιο λόγο να μιλήσουμε για την οικονομία των νέων. Αν υποστηρίξουμε την ε, πολιτική για τους νέους, θα καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω μια τέτοια εξέλιξη στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αν πετύχουμε ένα τέτοιο, μια τέτοια κίνηση, ένα τέτοιο, μια τέτοια βάση, θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε, στο μέλλον και άλλες σχετικές πολιτικές. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδίως μετά την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως έλεγε η εισηγήτρια, είναι γεγονός ότι ο προϋπολογισμός θα είναι μια δοκιμή, ένα πρώτο τεστ για το πώς θα λειτουργήσει ο προϋπολογισμός με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό θα ήθελα ε, σε αυτή την πρώτη δοκιμή να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία που μέχρι τώρα ακολουθήσαμε. Θα ήθελα λοιπόν να προσαρμόσουμε την εργασία μας εν ώψη της πρώτης ανάγνωσης της Κομισιόν και της Επιτροπής, ιδιαίτερα εν ώψη της συνδιαλλαγής του Νοεμβρίου διότι όντως τα προηγούμενα χρόνια, εγώ μόνο από την προηγούμενη χρονιά είχα, αλλά από ό,τι έμαθα, πάντα στις προηγούμενες συνδιαλλαγές ερχόντουσαν όλοι με 300, 400, 500 τροπολογίες, αλλά στην πράξη 15-20 μένανε. Θα μπορούσαμε να προλάβουμε την διαδικασία αυτή και εν τέλει οι τροπολογίες αυτές, η δουλειά που θα έχουμε επιτάπητος για να συζητήσουμε το Συμβούλιο, θα μπορούσε να γίνει με τρόπο ούτως ώστε να υπάρξει πραγματική συζήτηση στη συνδιαλλαγή των θεμάτων επί των οποίων θα υπάρχει πραγματική διαφορά και απόψεων και επί των οποίων θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Γι' αυτό θα έπρεπε λοιπόν από πλευρά μα να χτενίσουμε καλύτερα την προγενέστερη δουλειά πριν την ε, συνδιαλλαγή του Νοεμβρίου και γι' αυτό θα πρέπει να δοκιμάσουμε με πολλού τρόπου, πολλέ πρωτοβουλίε. Μεγαλύτερη προτεραιότητα στι εξειδικευμένε επιτροπέ. Να ζητήσουμε από τι επιτροπέ εκείνε, όπω έγινε στην Επιτροπή Προπολογισμών για παράδειγμα, να ασχολούνται πιο διεξοδικά, νωρίτερα και να έχουν περισσότερες επαφές μαζί μας από το ξεκίνημα. Το άλλο σημαντικό θέμα. Να ξεκινούμε νωρίτερα από τη στιγμή που έχουμε τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου ένα προσχέδιο προϋπολογισμού να συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το Συμβούλιο. Δίπλα-δίπλα. Πολύ νωρίτερα από αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα, ούτως ώστε να υπάρχει συντονισμός με το Συμβούλιο από τη στιγμή που έχουμε το σχέδιο προϋπολογισμού επιτάπητος. Αυτό μου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά για το πώς μπορεί να γίνει αυτός ο συντονισμός λέγοντας, βλέποντας ότι χάνεται η συνδιαλλαγή. Εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω στο χρονοδιάγραμμα συνδιαλλαγή τον Ιούλιο. Πώς θα γίνει ο συντονισμός αυτός. Εάν δεν γίνει με, το συντονισμό, με, με τη συνδιαλλαγή του Ιουλίου θα υπάρξουν άλλοι τρόποι. Αν δεν μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να συντονίσουμε τις εργασίες μας με το Συμβούλιο νωρίτερα, δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον συντονισμό αυτό. Κάτι άλλο που δεν εμφανίζεται στο κείμενο. Πρέπει να εξετάσουμε πώς ε, θα συσχετίσουμε την παρουσία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ή πώς θα δώσουμε κάποια εντολή στην εισηγήτρια κατά βάση εν ώψη των συνδιαλογών, των συναντήσεων, των τριμερών διαλόγων με το Συμβούλιο. Αυτά. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ, Ειντερ. Έκανα κάποιο λάθος, κάποια άκομψη παρατηρήση και αυτό ε, με οδήγησε στο να ζητήσουν πολλοί άντρε το λόγο. Ε, τους δίνω το λόγο, αλλά να είναι πολύ σύντομοι παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ο κύριος Γκουτμάνης. να πω στην εισηγήτρια. Υπάρχει πολύ καλή χρήση του υπολογισμού διότι φαντάζομαι ότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρουσιάσει κάτι καινούργιο ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις συνεχώς με παγιές τρόπους προσπαθούν να καλύψουν τα προβλήματα. Υποστηρίζω το σημείο 6 στη σελίδα 4 που είναι οι συνολικές επιπτώσεις του προϋπολογισμού. Έχω ήδη ετοιμάσει ένα κείμενο γραπτό, τελείως διαφορετικό από αυτό που περιλαμβάνεται μέχρι τώρα. Είσαστε πολύ αισιόδοξοι για την κατάσταση. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Εγώ αναφέρω ότι οι διαδικασίες ε, εκπλήρωσης είναι πολύ χαμηλές. Ζητούμε λοιπόν από την Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί για να μην έχουμε τα ίδια πράγματα με την προηγούμενη φάση της δημοσιονομικής προοπτικής όταν το Ταμείο Συνοχής ε, είχε εξαιρετικά μεγάλη υποκατανάλωση. Βέβαια, ε, μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα για εσάς, αλλά είναι το 30% του προϋπολογισμού της Ένωσης τα διαφορετικά ταμεία. Σας είπα ότι εγώ γενικά είμαι υπέρ του να υποστηρίζουμε θετικά πράγματα, αλλά μερικές φορές πρέπει να ε, έχουμε και μια πιο καλή εικόνα της πραγματικότητας. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο φαγητό μας ε, που μας ε, ετοιμάζει η συντόνια έχει λίγο αλάτι, λίγο ξύδι. Ο κύριος Σούριαν, να σας πω κάτι που μπορεί να σε εκπλήξει. Το ΕΛΚ υποστηρίζει την έκθεση και το σχέδιο γνωμοδότησης. Για την τελευταία παρατήρηση του συναδέλφου. Σωστά τα λέει. σκεφτόμουν την γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή. Ήμουνα εισηγητής και ίσως να υποβάλω και εγώ κανένα δύο τροπολογίες για το θέμα αυτό. Δεν είναι πολύ καλό το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Η συζήτηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης για τα Διευθυντικά Ταμεία θα γίνουν μέσα Μαρτίου, μετά την ολοκλήρωση δηλαδή αυτής της καθηγητήρια, αυτών των καθηγητήριων γραμμών, λαμβάνοντας τόσο υπόψη ότι τα στοιχεία από την Επιτροπή θα έρθουν νωρίτερα, και μπορεί να φανταστεί κανείς πως η κατάσταση τώρα, πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε δυναμικά μηνύματα ακριβώς όπως προναφέρθηκαν. Το μόνο θέμα που μου δημιουργεί κάποιες επιφυλάξεις είναι αν αναλύσουμε την κατάσταση στον τομέα των πληρωμών θα δείτε ότι είναι χάλια κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη. Σημαντικά καλύτερη η απόσταση μεταξύ ωστόσο υποχρεώσεων και πληρωμών, ο δρόμος μάλλον από τις υποχρεώσεις μέχρι τις πληρωμές, είναι δύσβατος. Και όταν έχεις μεγάλο ποσοστό δεσμεύσεων, δεν σημαίνει για καλά ότι θα υπάρξει πραγματική ανάλωση των χρημάτων. Λογικό λοιπόν είναι η Επιτροπή Προπολογισμών να ασχολείται κυρίως με πληρωμές. Το χρήσιμο τμήμα της πολιτικής συνοχής είναι αν τα λεφτά είναι στη χώρα και δουλεύουν εκεί, το να λέμε μόνο για σχέδια, τούτο αποτελεί προκαταρτικό μόνο βήμα. Μόνο όταν κατεβαίνουν τα λεφτά καταλαβαίνει ο κόσμος τα αποτελέσματα. Και όταν και εκεί στις πληρωμές υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Να ζητήσουμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν, ιδίω γιατί ζούμε μία φάση κρίσεως. Τα διαφορετικά ταμεία είναι ένα εργαλείο που, θα επιτρέ... που μπορεί να επιτρέψει στην Ένωση να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την κρίση. Αυτή ήταν η πολιτική και πέρσι και φέτος και πάντα. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους νέους. Η Ευρώπη είναι εδώ πάντα να σε σταθεί δίπλα όταν υπάρχει ανάγκη. Και τώρα υπάρχει ανάγκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Πόρτας. Ε, θα είμαι σύντομο, έλεγα. Ήθελα να πω ότι η κυρία Συντόνια έκανε, είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ωστόσο, κάποιο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω περισσότερο είναι, μίλησε για την έμφαση στις προτεραιότητες στους νέους, ε, για το πέρασμα από τις σπουδέ στη δουλειά, προσπαθώντας ακριβώς να συνδέσει καλύτερα την, ε, το πέρασμα από τις σπουδέ στη δουλειά και την ανάγκη να υπάρχει μια εγκάρσια προσέγγιση των διαφόρων προγραμμάτων με σημαντική ε, με συμβολή της Ένωσης. Ωστόσο, το πρόβλημα εδώ δεν ε, περιλαμβάνει μόνο, δεν, είναι με αυτόνομο, πρέπει να έχει σύνδεση και με την ευρύτερη πολιτική έρευνας. Μην ξεχνάτε το εξής, για ένα νέο ερευνητή, αυτό που του αλλάζει τη ζωή είναι το ότι σταματάει να είναι ε, σε μια επαγγελματική αβεβαιότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα ωστόσο τη ερευνητική κοινότητα στην Ευρώπη σήμερα. Γι' αυτό ο προπολογισμό δεν δίνει αποτελέσματα. Η απάντηση είναι πολύ χαμηλότερη, πολύ λιγότερο σημαντική από τις προσδοκίες. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να γνωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια προτεραιότητα που να έχει πολιτικό χαρακτήρα. Τα προγράμματα για τους νέους είναι αστεία σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού. Οποιαδήποτε αύξηση ποσοστιαία θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα λίγο φενάκι. Υπάρχουν βέβαια και οι πολιτικοί κίνδυνοι. Ωστόσο, είναι σημαντικό το ότι μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Επιπλέον, συμφωνώ με τη Γιούτα Χάουγκ. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε το θέμα της αλλαγής του κλίματος. Πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Προσαρμογής καλύτερα. Το κείμενο όπως έχει αυτή τη στιγμή δεν με ικανοποιεί θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε διότι η μόνιμη θεσμοποίηση ενός ε, συστήματος μόνιμης υποστήριξης τη ενίσχυση τιμών είναι συζητήσιμο. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην τιμή. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση να υιοθετήσουμε μια νέα προσέγγιση στον τομέα. Ένα τελευταίο θέμα, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε. Μπορείτε να μου διευκρινίσετε κάπως καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει στην αναθεώρηση, ε, στην ενδιάμεση αναθεώρηση των προοπτικών. Θα είναι ad Αναθεώρηση δεν θα αλλάζει δηλαδή τα μεγάλα κομμάτια του προπολογισμού ή όχι. Το περιθώριο χειρισμού για τον τωρινό και για τον μελλοντικό προπολογισμό είναι μικρά. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τις προοπτικές τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2015-2016 ουσιαστικά ή όχι, σημαίνει ότι θα, έχουμε, θα αλλάξουμε ριζικά την αντιμετώπιση του προπολογισμού. Αν θέλουμε κάτι τέτοιο, αν θέλουμε δηλαδή βασικέ αλλαγέ, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν με τον προπολογισμό και με διαφορετική προσέγγιση. Αλλιώ όμω είναι τα πράγματα αν δεν αλλάξουν ε, οι, βασικές, α, οι βασικοί άξονες της δημοσιονομικής πολιτικής. Ο κύριος Φέρμ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Τα σημαντικότερα ζητήματα έχουν καλυφθεί από τους συναδέλφου συναδέλφους μου. Θα ήθελα να αφαιρθώ λίγο στη διαδικασία. Καταρχάς να πω αυτό που είπε και η Αν Γένσεν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο για τη σύνθεση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής. Αφήστε τις πολιτικές ομάδες να αποφασίσουν. Δεύτερον, αυτό που πει Έντερ είναι πολύ σημαντικό. Η περίοδος εκείνη που μεσολαβεί ανάμεσα στην παρουσίαση του σχεδίου προπολογισμού αρχές Μαΐου και τι διακοπέ για το καλοκαίρι. Τότε ουσιαστικά μπορεί να ξεκινήσει ο διάλογος με το Συμβούλιο και τότε μπορούμε να διαμορφώσουμε την εντολή διαπραγματεύσή μα. Δεν έχουμε όμω πλέον τώρα τη συνδιαλλαγή του καλοκαιριού, έτσι δεν είναι. Μολονότι οι περισσότεροι από εσά μάλλον δεν τη θέλετε, μολονότι βέβαια ήταν χρήσιμη στο παρελθόν. Αυτό που μου λείπει όμω είναι η συζήτηση για την εντολή πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο για να συζητήσουμε τη δική μας εντολή. Αν θα έχουμε δηλαδή εντολή για τριμερή διάλογο ή για την Επιτροπή Συνδιαλλαγής ή για κάποιες άλλες συζητήσεις. Για δημοκρατικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα αυτή, να μπορούμε να συζητήσουμε δηλαδή την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι πολύ σημαντικό να εμπλέξουμε συζήτηση αυτή και τις άλλες επιτροπές στο στάδιο αυτό, προκειμένου να ανοίξει ο διάλογο με το Συμβούλιο πριν το καλοκαίρι. Δεν έχω να κάνω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις στη φάση αυτή. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή τη φάση της διαδικασίας και να μην αφήσουμε τα πάντα στα χέρια της Επιτροπής Συνδιαλλαγής. Θα πρέπει και η Επιτροπή Προπολογισμών να εμπλέκει τη διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν η Επιτροπή Συνδιαλλαγής και ο Τριμερής Διάλογος να λάβουν όλα τα ζητήματα. Επομένως, ζητώ από την η συγγήτρια και από τον πρόεδρο της Επιτροπής μας να σκεφτούν το ζήτημα αυτό. Τι θα κάνουμε δηλαδή με τα διαδικαστικά ζητήματα. Ενδεχομένως να πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο έγγραφο, κάποιο κείμενο, ένα ψήφισμα όπου θα συζητάμε την ε, εντολή μας, όχι τις μεγάλες προτεραιότητες όπως συζητάμε τώρα, αλλά να επικεντρωθούμε ακριβώς στο ζήτημα της ε, διαδικασίας επί του προπολογισμού. Και μια τρίτη παρατήρηση, πολύ σύντομα, πιστεύω ότι δεν συμπεριλαμβάνεται αυτό στο κείμενο, αλλά πρέπει να συζητήσουμε τη διοργάνωση της συζήτησης στην Ολομέλεια γιατί οι συζητήσεις στην Ολομέλεια, πέρα από τη διαλλαγή του καλοκαιριού, ήταν και αυτές εξίσου βαρετές. Πρέπει λοιπόν η συζήτηση να γίνει πιο ενδιαφέρουσα. Θα θυμάται, η ότι στις αρχές του 2000, όταν εγώ ήμουν εισηγητής για τον προπολογισμό, να προσπαθήσαμε να καλέσουμε διάφορους ε, συμμετέχοντες στη συζήτηση για τον προπολογισμό και καλύψαμε διάφορες κατηγορίες και την, το τμήμα 4 και καλέσαμε και διάφορους α, ε, επιτρόπους ε, να συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή. Επομένως, ας ξανασκεφτούμε πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε την όλη συζήτηση επί του προπολογισμού λίγο πιο ενδιαφέρουσα, προκειμένου να αποφύγουμε τις βαρετές συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Γκέραν. Νομίζω ότι έχεις ε, δίκιο. Όντως, χρειαζόμαστε μια εντολή, μια εντολή και διαφορετική από την εντολή εκείνη την οποία έχει το Συμβούλιο σε σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε μία έγκριση της πολιτικής θέσης Επιτροπής Προπολογισμών που θα εγκριθεί στη συνέχεια από την Ολομέλεια και αυτή θα είναι η διαπραγματευτική εντολή που θα έχει η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα πάμε και στη συνδιαλλαγή. Όντω έχουμε ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα αυτή τη φορά, μία μόνο ανάγνωση προβλέπεται. Δεν προβλέπεται η συνδιαλλαγή του Ιουλίου. Πάντως, προτού γίνει ο τριμερής διάλογος του Ιουνίου, θα πρέπει να έχουμε μια διαπραγματευτική θέση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανωθούμε, η εισηγήτρια θα μας πει ποια είναι η αποψή της, προκειμένου να καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως. Συντόνια, δεν ξέρω αν θα θέλεις να καταλήξει κάποια συμπεράσματα σύντομα για να περάσουμε και στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης. Έχεις το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω πολύ σύντομα στις παρατηρήσεις που γίνανε. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό αν είχα το χρόνο. Ωστόσο θα προσπαθήσω να σα απαντήσω σύντομα. Δύο συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην αντιμετώπιση του, των κλιματικών αλλαγών. Περιλαμβάνεται μία σχετική πρόταση στην παράγραφο 33 ενδεχομένως θέλετε να ενισχύσετε λίγο τα όσα λέγονται στην παράγραφο 33. Πάντως γίνεται νήξη στην παράγραφο αυτή. Λέμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την καταπολέμηση της αλλαγής ε, του κλίματος. Και λέω στην έκθεση ότι αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τώρα το έγγραφο εργασίας. Το έγγραφο εργασίας αποτελεί σημείο κίνησης για περαιτέρω συζητήσεις. Μετά την ανταλλαγή απόψεων που έγινε εδώ θα προσπαθήσω να συντάξω κάποιες νέες παραγράφους για τις δημοσιονομικές προοπτικές προκειμένου να συζητηθούν και αυτές μαζί με τις υπόλοιπες ε, τροπολογίες. Η κυρία Γένσεν έφυγε από την αίθουσα, πάντως αναφέρθηκε και αυτή και άλλοι συνάδελφοι στην σύνθεση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε μία ανοιχτή προσέγγιση και να διευρύνουμε τη σύνθεσή μας προκειμένου να έχουμε και οι δήμονες στα πλαίσια της ομάδος μας. Δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο από τις προτάσεις που κάνω στο έγγραφο εργασία Πάντω, συμφωνώ με όσου είπαν ότι ενδεχομένω να είναι πολύ νωρί αυτή τη στιγμή για να αποφανθούμε για την οριστική σύνθεση τη αντιπροσωπεία μα στην Επιτροπή Συνδιαλλαγή. Αναφέρθηκα στι κλιματικέ αλλαγέ, οικονομία των νέων. Όσον αφορά τα σχόλια της κυρίας Καρδιαμπάλα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις α, τροπολογίες προτού πάμε στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή πως θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι έχουμε πλέον μία μόνο ανάγνωση και πως θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα έχοντας τόσες πολλές τροπολογίες, πολύ περισσότερες από τις προηγούμενες φορές. Είναι μία πρόκληση λοιπόν αυτή και χρειάζομαι και τη βοήθεια και των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων για να δούμε πως θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την περίπλοκη αυτή κατάσταση. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο τριμερής διάλογος και οι προετοιμασίες για τον τριμερή διάλογο του Ιουνίου έχουν προετοιμαστεί σωστά, ότι έχουμε χρόνο προκειμένου να καταφέρουμε να πάμε με μια ισχυρή θέση για το σχέδιο προπολογισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι σίγουρα τον Ιούνιο θα χρειαστεί να εργαστούμε πολύ. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε είχε να κάνει με τα παραδοσιακά στρατηγικά ζητήματα τα οποία πάντα συζητούσαμε στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προπολογισμού. Γνωρίζω τα ζητήματα αυτά, διαρθρωτικές πολιτικές, ουσιαστικά η κοινή γεωργική πολιτική. Τα ζητήματα αυτά δεν με βρίσκουν αδιάφοροι καθόλου. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα και γνωρίζω ότι αντιστοιχούν σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του προπολογισμού. Γνωρίζω επίσης ε, για τις σχετικές προκλήσεις και ενδεχομένως ορισμένα από τα παραδοσιακά εργαλεία που έχουμε για τους τομείς αυτούς να ξαναχρησιμοποιηθούν Πάντως, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τη συζήτηση για την εφαρμογή των διατροτικών πολιτικών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε εκ νέου τη συζήτηση και τον προπολογισμό και σε άλλους τομείς, έχοντας βέβαια πάντα κατά ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή εφαρμογή των όσων έχουμε αποφασίσει πολιτικά στο παρελθόν. Τώρα, όσον αφορά το τι συνέχεια θα δοθεί, το πώς θα καταφέρω ουσιαστικά να πραγματοποιήσω στην πράξη τις προτεραιότητές μου. Θα σας δώσω στο μέλλον ένα έγγραφο εργασίας όσον αφορά τα μέσα πολιτικής για τους νέους που έχουμε στα χέρια μας. Στις αρχές της Άνοιξης θα έχετε ένα τέτοιο έγγραφο εργασίας και σε αυτό το έγγραφο θα ήθελα να εμβαθύνω περισσότερο στα τι γίνεται, στο τι γίνεται στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού για τους νέους, ποια είναι τα προγράμματα για τους νέους, ποια είναι τα πιλωτικά προγράμματα που υφίστανται, αν όντω υπάρχουν προτάσεις ανάλογες με αυτές που έκανε ο κύριος Πόρτας, όσον αφορά δηλαδή την έρευνα, τους ερευνητές, την κινητικότητα των ερευνητών, τι γίνεται με τους νέους ερευνητές. Και στο έγγραφο εργασίας αναφέρομαι και στην πέμπτη αυτή ελευθερία, την κινητικότητα της ε, γνώσης. Για μένα όλα αυτά τα ζητήματα αλληλοσυνδέονται, επομένως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Κατέγραψα τις ε, παρατηρήσεις που κάνατε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Πολλά από αυτά θα συμπεριληφθούν ως ε, δικές σας δικές μου στις, ε, στην έκθεση που θα γίνει για τις ε, προτεραιότητες του προπολογισμού και πολλά από τα σχόλια αυτά επίσης θα τα δούμε και στα έγγραφα εργασίας τα οποία θα υποβάλουμε στο μέλλον και ιδίως στο έγγραφο αυτό εργασίας το οποίο θα αναφέρεται στα μέσα τα οποία διαθέτουμε για την πολιτική για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όσοι είπανε θετικά λόγια, θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα πρέπει να είστε πάρα πολύ ενθουσιώδης αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ο ενθουσιασμός να είναι ο ίδιος και, στο τέλος της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε συντόνια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μου κάνει εντύπωση και αυτό είναι πολύ θετικό. Μου κάνει εντύπωση αυτή η πολύ μεγάλη συνένεση που υπάρχει για την πολιτική για τους νέους, να δοθεί προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό είναι ένας ε, τομέας στον οποίο η ορατότητα στην οποία αναφερόμαστε για τις δράσεις Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να δείξουμε στους νέους που υποφελούνται από δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η χρηματοδότηση αυτή έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το λέω όχι για να σας αποθαρρύνω, αλλά για να συμπληρώσω τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν να σας υπενθυμίσω ότι η συντονία μαζί με τον ε, Λάζλου Σούριαν αναφέρθηκαν σε αυτό το έγγραφο εργασίας το οποίο αναφέρεται στα διαδικαστικά προβλήματα και το κάναμε αυτό γιατί μας το ζήτησε αυτό η διάσκεψη των Προέδρων. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου έστειλε μία επιστολή πριν από μερικέ εβδομάδε εξ ονόματο τη διάσκεψη των Προέδρων, ζητώντα από την Επιτροπή Προπολογισμών, και λέω στα αγγλικά, να υποβάλει στην Επιτροπή των, στην διάσκεψη των Προέδρων, μετά από συζήτηση με την διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, ένα έγγραφο εργασία για το ποιε θα είναι επιπτώσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα στην ετήσια διαδικασία κατάρτιση του προπολογισμού. Ιδίως όσον αφορά το νέο χρονοδιάγραμμα και ιδίως όσον αφορά την διοργανική προετοιμασία των ε, τελευταίων φάσεων της ε, ετήσια διαδικασίας κατάρτισης του προπολογισμού. Το καλύτερο λοιπόν θα ήταν να συμπεριλάβουμε τις απόψεις μας στην έκθεση που θα προετοιμάσει η Συντόνια και σε υπενθυμίζω το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση αυτή, όπως έκανε και η Συντόνια πριν από λίγο. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 25η Φεβρουαρίου στις 6. Ε, το Μάρτιο θα εγκρίνουμε την έκθεση στις 4 Μαρτίου και στην δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου θα εγκριθεί, θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή από, τον, από την ολομέλεια. Είναι σημαντική έκθεση αυτή γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγγράψει στη δική της σε διάταξη το ζήτημα αυτό, συγκεκριμένα σε μια συνεδρίαση που θα γίνει στις 11 Μαρτίου, επομένως θα μπορούσε και αυτή να εμπνευστεί, αν θέλετε, από την ψηφοφορία που θα γίνει εδώ στην Επιτροπή μας στις 4 ε, Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Σας προτείνω να περάσουμε τώρα στο σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο μπορούμε να καλύψουμε πολύ γρήγορα. Έχουμε εδώ μια έκθεση της Γιούτα Χάουγκ. Γιούτα, έχει το λόγο. Ja, danke. Ähm, der ist zwar wichtig, aber ich hoffe doch... Λοιπόν, ε, ναι. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μπορούμε να τελειώσουμε γρήγορα το θέμα αυτό. Πρόκειται γιατί τροποποίηση της αρχής εποπτείας, supervisory authority, εδώ και πολύ καιρό ζητάμε μια που έχει αλλάξει η βάση για την επιτροπή αυτή που εποπτείας για το κοριό κλπ. Και η Κομισιόν ανέλαβε την εφαρμογή του προγράμματος από τότε δηλαδή που ανέλαβε η Κομισιόν δεν είχε αυτή η Επιτροπή, η Αρχή Εποπτείας μια βάση εργασίας. Τώρα προτείνει η Κομισιόν μια αλλαγή. Καταρχήν δεν θα λέγεται αρχή αυτό πια, γιατί είναι υπερβολικό να το πούμε αρχή. Θα λέγεται υπηρεσία. Καλό είναι αυτό. Αυτή η agency, η υπηρεσία αυτή, λέει ότι είναι αρμόδια για την ε, έγκριση, για την ασφάλεια. Ωραίο αυτό. Εγώ υπέβαλα τροπολογίες εδώ, μία για το λεγόμενο νομοθετικό ψήφισμα, όπου αναφερόμαστε για άλλη μια φορά στο ότι χρειάζεται να υπάρχει συνεννόηση με το άλλο σκελό τη Δημοσιονομική Αρχή βάσει του άρθρου 47 όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη νέα αυτή υπηρεσία. Ένα αυτό. Μετά υπάρχουν τέσσερι τροπολογίε. Μία από αρά το άρθρο 47 πάλι. Και το θέμα της του προγραμματισμού του δημοσιονομικού προγραμματισμού για να μπορούσαν όλα αυτά να ενταχθούν μέσα στον προπολογισμό μα. Πρόκειται για τροπολογίε που γνωρίζετε πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και πολύ καιρό. Είναι οι συνήθειε μα τροπολογίε όταν πρόκειται για την ε, ίδρυση νέων υπηρεσιών ή την τροποποίηση παλιών. Δύο στοιχεία είναι καινούργια. Καταρχήν, ότι λέω κάτι όσον αφορά την διάρκεια της εντολής του Προέδρου, του, του Διευθυντή. Η Κομισιόν είχε πει έχουν αλλάξει γενικά η πολιτική της υπηρεσίας αυτές και τώρα αλλάζει η διάρκεια της θητείας αυτής από 5 στα 4 χρόνια. Αυτό δεν το είχαμε πει ποτέ όμως. Έχουμε γι' αυτό μια διαθεσμική ομάδα εργασίας. και εκείνοι που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ομάδα εργασία αυτή έχουν καθοριστεί και για την τρεξοθυσία. Την περασμένη εβδομάδα ο Παρόζο υποσχέθηκε σε μια συνάντηση όλων των υπηρεσιών ότι θα ορίσει σύντομα και του συναδέλφου από την Κομισιόν που θα συνεργάζονται στην Επιτροπή αυτή και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το θα προστίθε και η εκάστοτε Προεδρία του Συμβουλίου. Και εκεί θα εξεταστεί και το θέμα της ε, διάρκειας της θητείας των ε, διευθυντών. Αλλά όλα θα πρέπει να προσαρμοστούν για όλες τις υπηρεσίες, ομοιόμορφα. Εγώ θα υποβάλω την τροπολογία ότι και για αυτή την υπηρεσία, όπως και για όλες τις άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει να παραμείνουμε στην πενταετή θητεία του διευθυντή. Η τελευταία τροπολογία είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα. Εκεί προσπαθώ με την βοήθειά σας να ορίσω ότι η έδρα της υπηρεσίας θα παραμείνουν οι Βρυξέλλες. Έχουν αρχίσει τις εργασίες τους. Έχουν αρχίσει τις εργασίες τους εδώ, στις Βρυξέλλες. Λογικό είναι αυτό. Να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Αυτό μας στοιχίζει το λιγότερο τον ευρωπαϊκό προβλησμό δηλαδή. Και λέω ξεκάθαρα ότι ακόμα και αν πρόκειται για μια νέα υπηρεσία, θεωρούμε ότι θα πρέπει η έδρα της να είναι Βρυξέλλες. Αυτά. Τελεία και Παύλο. Ευχαριστώ, Γιούτα, για την παρουσίαση αυτή. Θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε την ε, άποψή μας για το νομικό σύστημα που διέπει την ε, εποπτεία του Γαλιλαίου. Η περασμένη επιτροπή είχε βρει τη δυνατότητα μιας λύσης για ένα θέμα που διέρε το κράτη-μέλη, δηλαδή την χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού Γαλιλαίου και είχαμε αποφασίσει να δώσουμε το σύνολο των οικονομίσεων που μπορούν να γίνουν στον προϋπολογισμό ΦΕΟΓΑ 2007 στη χρηματοδότηση του συνόλου του προγράμματος Καλλιλέο. Όπως προβλέπτω τότε υπάρχει ο κίνδυνο ότι το επίπεδο δαπανών αυτό θα ξεπεραστεί τους επόμενους, τα επόμενα χρόνια. Δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί. Αυτή τη στιγμή ε, τροποποιούμε την οργάνωση της εποπτείας, όπως το εξήγησε και η Γιούτα. Η Επιτροπή Ήτρε είναι υψουσία αρμόδια. Προθεσμία για τις τροπολογίες ορίζεται στις 26 Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα, 4 Μαρτίου δηλαδή, η ΙΤΡΕ θα ψηφίσει στις 17 και στην πρώτη σύνοδο του Απριλίου θα ψηφιστεί το θέμα στην Ολομέλεια. Λοιπόν, προτείνω τώρα να περάσουμε στα σημεία που θα ακολουθήσουν ψηφοφορίες, για να είμαστε σίγουροι ότι θα ψηφίσουμε ότι είναι στιγμή που προβλέπετε. Για τα σημαντικά σημεία για τα οποία όμως έχουμε ήδη ακούσει τις παρουσιάσεις και έχουμε κάνει τη συζήτηση στις προηγούμενες συνεδριάσεις και μπορούμε να πράσουμε μέσα στην ψηφοφορία. Έχουμε καταρχήν τρία σημεία που αφορούν την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ο εισηγητής ε, Ράμερ Μπέγκερ δεν μπορούσε να είναι παρόν, αλλά μα είχε προ... υποβάλει τι προτάσει του στην προηγούμενη συνεδρίαση και μπορούμε να περάσουμε μέσα στην ψηφοφορία, γνωρίζοντα ότι πάμε τροπολογίε. Prendre... Λοιπόν, θα εξετάσουμε το σημείο 14 καταρχήν. Κινητοποίηση του ταμείου αυτού ενίσχυση για την ε, παγκοσμιοποίηση για τη Λιθουανία.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 Α, όχι, όχι, για το 14 δεν υπάρχουν τροπολογίες όπως ξέρω. Αφορά τη Λιθουανία, το σημείο 14, χωρίς τροπολογίες. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Απουσία του. Σας το παρουσιάζω. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Αν κρίνεται. Με ευρία πλειοψηφία. Περνάμε τώρα στο σημείο 12. Το απόβληση του ίδιου ταμείου για τους γερμανούς εργαζόμενους που έχουν απολυθεί στα πλαίσια της αναδιόρθρωσης, αναδιοργάνωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και εδώ έχουμε μία τροπολογία του συναδέλφου Αλβάρο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Είναι κάπως ατυχές ότι εγκρίναμε την πρώτη. Γιατί η δική μου προφορική τροπολογία αφορά και τις τρεις εκθέσεις του συναδέλφου Μπέγκε. Γιατί και στις τρεις υπάρχει διατύπωση, στα αγγλικά υπάρχει εδώ, τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όσοι δυνατότητες για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ε, παγκόσμια οικονομικής και χρηματοπιστής ε, κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό τους ε, ρόλο κλπ. Η πρότασή μου είναι μετά το άνοκο να αλλάξουμε τον τονισμό που αποδίδουμε στο ταμείο αυτό και αυτό για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτά. Pardon. Euh, oui, euh, pardon mon cher collègue, donc Συγγνώμη, συνάδελφε. Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται και για τη Θα ψηφίσουμε λοιπόν αναδρομικά το Ποτινά. Γιατί πρόκειται για μια τροπολογία που αφορά και τις τρεις προτάσεις ενίσχυσης. Νόμιζα ότι δεν υπήρχε για την... Ε, δεν υπήρχε έτοιμα τροπολογίας για τις προηγούμενες δύο προτάσεις, αλλά μόνο για την Λιθουανία. Πάντω ισχύει και για τι τρει. Ο Ράιμον Μπέγκε δεν είναι υπέρ, αλλά ο Σαλβαδόρ που ήρθε και τον οποίο καλωσορίζουμε, ήρθε καθυστερημένα, λόγω ενός σπάνιου γεγονότο φαινομένου στη Γαλλία, μια απεργία. Όταν στη Γαλλία υπάρχει, γίνεται απεργία, τα αεροπλάνα που έρχονται από την Ισπανία και προσγειώνται στι Βρυξέλλε πρέπει να περάσουν από πιο γαλήνιους ουρανούς. Πρέπει να γνωρίζει ότι η απεργία αυτή είναι μια απεργία κατά του ε, open sky, του ενιαίου ουρανού, του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πτήσεων. Ορισμένοι Γάλλοι εργαζόμενοι θέλουν τα σύνορα που καταργήθηκαν από το 1993 ήδη για τα χερσαία σύνορα της χώρας, των χωρών μας να συνεχίσουν να υφίστανται μεταξύ των νεφών. Χαιρόμαστε πάντως που κατάφερε και ήρθε παρόλα αυτά ο Σαλβαδόρ μαζί του. Η ομάδα του μας είπε ότι είναι κατά, ψηφίζουμε την τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας Αλβαρό που αφορά και τις τρεις προτάσεις. Μετράμε. 17, 8, 9, 10, 11, 12. 13-14 même. 13-14. Qui est contre κατά. Une majorité favorable. Η πλειοψηφία είναι υπέρ. Συγχαίρουμε τον κύριο Άλβαρο. Α, αργήσατε, αργήσατε, αργήσατε. Δεν αλλάζει τίποτα όμως. Έρχεται τρέχοντας η Μπάρμπαρα να καταψηφίσει τον Άλβαρο, δεν ξέρω τι έχετε μεταξύ σας. Τέλος πάντων, ο Άλβαρο κέρδισε. Και αφορά και τις τρεις προτάσεις. Προχωρούμε. Για το σημείο 12 κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση των, των εργαζομένων στην ε, αυτοκινητοποιημένη τη Γερμανία. Ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ είμαστε, φαντάζομαι. Κατά. Και ένας είναι κατά. Αποχές. Μία αποχή. Συνεχίζουμε. Σημείο 13. Στον κλάδο των ψυγείων. Η ίδια κινητοποίηση. Για ποια χώρα είναι αυτή τα ψυγεία? c'est la Lituanie aussi, non Oui, c'est Lituanie aussi. Πάλι για τη Λιθουανία. Τα ψυγεία στην Λιθουανία. Ε, κατά, τη, κατά βάση στη χώρα αυτή, για το μεγαλύτερο τμήμα του έτου. δεν χρειάζονται ψυγεία, αλλά τέλο πάντων. Ποιοι είναι υπέρ τη δράση αυτή των εργαζομένων που φτιάχνουν το χειμώνα ψυγεία στη Λιθουανία. Κατά, αποχές, δεν υπάρχουν αποχές. Δεκτό Ομόφωνο με τις τρεις τοπολογίες του κύριου Άλβαρο. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε τις, τη μετακίνηση, τη μεταφορά των πιστώσεων. Κύριος Σούριαν Νούμερο... euh, c'est le point numéro 16. Donc Το σημείο 16. Προτείνω να ψηφίσουμε από κοινού τρεις μεταφορές για τις τρεις δράσεις για τις οποίες είπαμε καταρχήν οκ. Okay. Ποιοι είναι υπέρ της μεταφοράς. Κατά. Αποχές. Η συντόνια είναι και υπέρ και κατά και απέχει. Εγκρίνεται το σημείο αυτό. Συγχαίρω τον εισηγητή και ευχαριστώ την Επιτροπή μας. Έχουμε να ψηφίσουμε και δύο ακόμα σημεία. Πρώτον, να ψηφίσουμε μια έκθεση του κυρίου Ντεάν για μια μικρή τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού του ακαθαρίστου εθνικού εισοδήματος. Ενό θέματο που μέχρι πρόσφατα μπορούσε να θεωρηθεί ω αποκλειστικά τεχνικό, αλλά οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν ορισμένα μέλη της ζώνης ευρώ δείχνουν ότι δεν είναι μόνο τεχνικά τα θέματα. Ζαν Λουικ, παρακαλώ. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. έγινε μία συζήτηση σε προηγούμενη συνάντηση. Δύο τροπολογίες ε, έχουν στόχο να ευθυγραμμίσουν το κείμενο στα γνωστά πλέον συμπεράσματα του Συμβουλίου. Προτείνω να υπερψηφίσουμε τις δύο αυτές τροπολογίες. Ευχαριστώ, Ζανλουίκ. Δείτε από για τις συνέπειες ότι αφορά τη συνεισφορά των χωρών σας στον κοινωτικό προπολογισμό δεν είναι αμεληταίο. Γιατί η Γαλλία μειώνει, τυχαίο είναι εγώ δεν φταίω, κατά 160 εκατομμύρια τη συνεισφορά τη Γαλλίας στον κοινωτικό προπολογισμό. 170 εκατομμύρια. 170 εκατομμύρια στα 18 δις περίπου. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης αυτής του κυρίου Ντέαν. Με τις δύο, α, υπάρχουν δύο τοπολογίες, όχι, όχι, όχι να ψηφίσουμε κάθε τροπολογία ξεχωριστά. Πρώτη τροπολογία. Κατάργηση, κακοί είμαστε, του άρθρου 2. Προτείνει ο εισηγητής. Υπέρ της κακή αυτή, της κακόπιστη αυτή τροπολογία του εισηγητή. Κατά αποχές κανείς δεκτό το κείμενο. Τροπολογία 2 που έχει ως στόχο να αναβάλει την εφαρμογή να στην ουσία αρνείται την αναδρομικότητα. Δηλαδή ο υπολογισμός αυτός δεν εφαρμόζεται αναδρομικά από την πρώτη πρώτου του 7 αλλά από την πρώτη πρώτου του 10. Τώρα δηλαδή. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Κανείς. Εγκρίνει το μόφωνο. Υπέρ της έκθεσης συνολικά του κύριου Ντεάν. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Έχουμε τώρα κάποιες μεταφορές του Λάζλο και κάποιες του κυρίου Μάνκα. Τώρα να δούμε πρώτα τις μεταφορές για την Επιτροπή 2010. Τρεις υπάρχουν. Δεκ, θα πει Δεκέμβριο δεκ. Όχι. Το ΔΕΚ έχει πολλά αρχικά στα γαλλικά. Το δεκ 01. Απόφαση σημαίνει. δεκ decision. Απόφαση 1. Γάλα. Χρησιμοποίηση των γαλακτοκομικών πόρων. Επιτέλους. Λάζλο.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 να βοηθά δηλαδή την γαλακτοκομική παραγωγή με 300 εκατομμύρια. Πολύ ωραία. Άρα δεχόμαστε την μεταφορά, έρουμε, το βγάζουμε από το αποθεματικό εφόσον η Επιτροπή, από τη στιγμή μάλλον που η Επιτροπή πρότεινε να ε, περάσει το άρθρο 186, να εφαρμοστεί το άρθρο 186 στον γαλακτοκομικό τομέα όπως το ζητήσαμε. Ποιοι είναι υπέρ μεταφοράς αυτής. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. ΔΕΚ 07. Διοικητικές δαπάνες. Κύριε Σιγητά. Ε, στο σημείο αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε απλά και μόνο. Έχω ορισμένε ερωτήσει. Ελπίζω να μπορέσει να απαντήσει η Επιτροπή. Πρώτον, τελειώνει περίπου ο Φεβρουάριο, αλλά είμαστε στο ξεκίνημα του έτους. Βλέποντας γιατί βλέπω ότι είναι λογικές οι δράσεις αυτές, αλλά ήταν γνωστές ε, όταν ε, ξεκίνησε η διαμόρφωση του σχεδίου προπολογισμού. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αυτές οι προτάσεις δεν είχαν συμπεριληφθεί στον προπολογισμό που ψηφίσαμε το Δεκέμβριο. Αναφέρεται για παράδειγμα η Ισλανδία εν ώψη της διεύρυνσης. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλουν κάποιες επιπλέον θέσεις. Μπορώ να δεχθώ ότι είναι προσωρινή ε, ότι τέλο πάντων ε, δεν είναι μόνιμε οι θέσει, αλλά είναι προσωρινέ. Αλλά αυτό ξεκίνησε από το καλοκαίρι. Το ξέραμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, ρωτώ, γιατί δεν μπήκε στην κανονική διαδικασία και απαιτείται με μεταφορά πιστώσεων. Η μεταφορά αυτή έχει τρία κομμάτια. Το ένα, το δεύτερο είναι η Ισλανδία. Το άλλο αφορά θέσεις εργασίας που έχουν παγώσει και έχουν πάψει και θα πάψουν να υπάρχουν το 2011. Γιατί καλύπτουμε αυτές τις παγωμένες θέσεις με έκτακτους υπαλλήλους. Το μυαλό μου φαίνεται δεν είναι αρκετά έξυπνο για το καταλάβει. Στον προπολογισμό εμείς ζητήσαμε να υπάρχει μια γραμμή αποθεματικού που θα διαχειρίζεται απρόβλεπτα προβλήματα κατά τη διάρκεια του έτους που απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό για νέες θέσεις. Ως κοινοβούλιο Λέμε ευελιξία, ευελιξία, ευελιξία. Ψηφίζουμε τα κονδύλια αυτά για το σκοπό αυτό, όπως είναι σαφές και από, την, ε, και από το σχόλιο. Ε, έχω μια, ε, κάποια ερωτηματικά. Δεν είμαι κατά. Ρωτώ. Ξέρετε τις ανάγκες αυτές και πριν ξεκινήσει ο προπολογισμό. Μήπως αυτή η καθυστέρηση είναι μια πράξη αυροφροσύνης προς τη νέα επιτροπή. Δηλαδή η παλιά επιτροπή δεν ήθελε να αποφασίσει για ένα θέμα που θα εφαρμόσει η νέα επιτροπή. Αυτή είναι μία εξήγηση που φαντάζομαι ότι είναι αληθινή. Δεν το ξέρω όμως. Μήπως μπορεί να μας εξηγήσει λοιπόν η Επιτροπή γιατί αυτή η ανάγκη μεταφοράς τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μόλις μου απαντήσουν θα σας πω τι προτείνω. Ευχαριστούμε. Είναι εδώ ο κύριος Γενικός Διευθυντής. Μπορεί να ξεκαθαρίσει λίγο τον εγκέφαλο του συναδέλφου, εισηγητού. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω κάπως το μυαλό του κυρίου Σούριαν να υπενθυμίσω μια βασική αρχή. Δεν μιλάμε εδώ για διορθωτικό προπολογισμό, μιλάμε απλώς για μια μεταφορά πιστώσεων. Δεν αλλάζουν λοιπόν τα ποσά, τα σφαιρικά ποσά δεν τροποποιούνται. Πρώτον αυτόν, δεύτερον. Όσον αφορά το ζήτημα της Ισλανδίας, να σα υπενθυμίσω κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το χρονοδιάγραμμα. Στα πλαίσια της καρτάρτης του προπολογισμού κάναμε μια πρόταση για το 2010 όσον αφορά τους σχετικούς πόρους και όταν εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο το προσχέδιο του προπολογισμού, τον Απρίλιο του 2009, η προπτική μιας προσχώρησης ή μιας ενδεχόμενης διαδικασίας προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, προβλεπόταν καθόλου σε εκείνη τη φάση. Θα θυμάστε ότι το Συμβούλιο συμφώνησε να γνωμοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 ε, Ιουλίου του 2009. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια συγκεκριμένη μονάδα τον Σεπτέμβριο του 2009, προκειμένου να προετοιμάσει τις απαραίτητες εργασίες που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο τέλος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να κινητοποιηθούν κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι αποσπάστηκαν από άλλες μονάδες Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να καταφέρουν να ασχοληθούν αμέσως με το ζήτημα αυτό. Η πρότασή μας λοιπόν έγινε τότε ζητούσαμε να γίνει μία προσαρμογή προκειμένου να αποζημιώσουμε τις μονάδες αυτές για τα άτομα εκείνα τα οποία έπρεπε να φύγουν από τα συγκεκριμένα τμήματα και να πάνε στην ειδική ομάδα εργασίας για την Ισλανδία προκειμένου να μπορέσουν δηλαδή να συνεχίσουν την φυσιολογική τους δουλειά και οι υπόλοιπε μονάδες, τα υπόλοιπα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι μια πολύ απλή εξήγηση λοιπόν. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Σούριαν, Έγινε εδώ πέρα μία μετάβαση από, το, από την κατηγορία ΔΕΛΤΑ, η οποία θα καταργηθεί, D, σε προσωρινούς ε, συμβασιούχους, ουσιαστικά. 14 είναι οι συμβασιούχοι αυτοί, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους υπαλλήλους του, της κατηγορίας ΔΕΛΤΑ, D, και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να αποζημίωσουμε ουσιαστικά, προσπαθήσαμε να αντισταθμίσουμε με τους συμβουλεσιούχους αυτούς τις κατηγορίες εκείνες, τις, μάλλον τα πόστα εκείνα της κατηγορίας Δέλτα, τα οποία θα εξαφανιστούν πλέον από τον κατάλογο των ανθρωπίνων πόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έρχεται αυτό σε συνέχεια της μεταρρύθμισης που έγινε για το καταστατικό του προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2004 και κατά αυτόν τον τρόπο η, προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα ε, την πολιτική προσλήψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να μην έχει έντονες οικονομικές επιπτώσεις, να μην αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε εξωτερικούς φορείς. Αυτά είχα να πω απάντηση προς τον κύριο Σούριαν και είμαι στην διάθεσή του προφανώς για περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά. Κύριε εισηγητή έχετε ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις αυτές. Ναι, πολύ ωραία. Επομένως μπορούμε να υπερψηφίσουμε. Πολύ ωραία. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής των πιστώσεων, κατά, Αποχές. Μία. Αποχή. Εγκρίνεται. Μία τελευταία φορά μετα... μεταφορά πιστώσεων πρέπει να εξετάσουμε. Ενημερωθήκαμε για αυτήν χθε. Απόφαση 08. Ε, μεταφορά πιστώσεων για την ΑΕΤ. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν είπαμε ότι σε περίπτωση επίγουσας ανάγκης είμαστε πάρα πολύ αργοί. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ ικανοποιημένο που μπορούμε να πούμε ναι για τη μεταφορά αυτή πιστώσεων. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, ποιο θα σηκώσει γρήγορα το χέρι για να βοηθήσουμε την IT. Σας ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Καμία. Επομένως, ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι αυτή τη, φορά στη μεταφορά πιστώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως δεν είχε ιδιαίτερη ορατότητα, δεν ήταν πάρα πολύ εμφανή στη δράση της για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτή στην ΑΕΤ. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να διορθώσουμε έστω και αργά λίγο την κατάσταση. Ευχαριστούμε τον κύριο Σουριάν. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιες μεταφορές πιστώσεων για τα άλλα θεσμικά όργανα. Ο κύριος Μάνκα μία μόνο μεταφορά, λέει ο Πρόεδρος, που έχει να κάνει με, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από τη στιγμή που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η συνθήκη της Λισαβόνα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έπρεπε να τηρήσει το άρθρο 50 των διατάξεων όσον αφορά την προσωρινή συνταξιοδότηση, την πρόορη συνταξιοδότηση. Προτείνω λοιπόν υπέρ της μεταφοράς των πιστώσεων αυτών. Σας ευχαριστούμε. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής πιστώσεων, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία και μπορούμε λέει ο Πρόεδρος, μάλλον υπάρχει μια συζήτηση πρέπει να γίνει για τις κατευθυντήριες ε, γραμμές. Από την άλλη όμως θα έχουμε μαζί μας και τον Γενικό Γραμματέα. Ας περιμένουμε λοιπόν λίγα λεπτά και ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκότμανης, ο οποίος ε, μας ζήτησε λίγο χρόνο προκειμένου να μας παρουσιάσει πολύ γρήγορα κινηματογραφικά σε άμεση σύνδεση με το Hollywood μία έκθεση που έχει να κάνει με ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κύριε Γκοτμανής, έχετε το λόγο. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά παίρνω το λόγο. Έχω προετοιμάσει την ομιλία μου, τώρα ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι δεν μπορεί να τη διαβάσετε από την οθόνη. Παρ' όλα αυτά, ας δούμε κάποιους πίνακες. Τι είναι αυτοί οι πίνακες. Πίνακες των διαφροντικών ταμείων του Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Ο λόγος για τον οποίο δεν σας έδωσα τους πίνακες αυτούς ε, σε έγγραφο είναι επειδή πρέπει να τους ελέγξω πρώτα. Τους υπέβαλα μόνο στον πρόεδρό μας και στη Γενική Διεύθυνση Ρέτζι. Έκανα ο ίδιος κάποιους υπολογισμούς και τα δεδομένα αυτά δεν είναι απόλυτα επαληθευμένα. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, μπορώ να σας πω ότι η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Οι πληρωμές, που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προς τα κράτη-μέλη και δεν αναφέρομαι εδώ πέρα στους εθνικούς προπολογισμούς, αναφέρομαι σε πληρωμές για την περίοδο 2007-2013, αν πάρετε το σύνολο των ταμείων, είναι μόνο 8%, 8,6%. Αυτό είναι το μέσο ποσοστό το οποίο προκύπτει. Και βρισκόμαστε στο τέλος της περίοδου των τεσσάρων ετών και δεν πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους αρχικούς μας στόχους. Και το πιο προβληματικό ζήτημα είναι ότι ε, έχουμε ολοκληρώσει την ε, χρηματοδοτική περίοδο 2000 μέχρι 2006 και 1,5 εκατομμύρια δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο κοινοτικό ταμείο και 1,2 εκατομμύρια για το Ταμείο Συνοχής. 2 εκατομμύρια, 2 δισεκατομμύρια έχουν χαθεί ουσιαστικά από την αρχική ανάληψη υποχρεώσεων. Και κάτι ακόμα. Το 8,6% είναι ο μέσος όρος. Το 63% των κρατών μελών βρίσκονται κάτω από το ποσοστό αυτό και ορισμένα βρίσκονται μόνο στο 3%. Το καλύτερο ποσοστό είναι 17,2%. Αν δείτε το σύνολο λοιπόν των ταμείων, η αρχική κατάσταση είναι ότι τα κράτη-μέλη με τα τη μεγαλύτερη, την μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων από την ευρωπαϊκή κοινότητα έχουν μεγαλύτερα ποσοστά απορρόφησης. Ουσιαστικά αναφέρομαι σε χώρες που φτάνουν στο ποσοστό του 300% καταφέρνουν να καλύψουν τα, να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αυτούς κατά 10, 12 ή ακόμα και 17%. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένε ε, χώρες. Από την άλλη έχουμε και άλλες χώρες όπου έχουμε πολύ μικρή αποστολή χρηματοδο... μάλλον πολύ μικρή χρηματοδότηση κατά κεφαλή και οι χώρες αυτές δεν έχουν καλή απορρόφηση. Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τα στοιχεία για ΑΕΠ, ούτε με το δημόσιο έλλειμμα των κρατών αυτών. Είναι εντελώς άσχετα πράγματα αυτά. Και τι βλέπουμε στο τέλος. Σας έδωσα κάποια γενικά στοιχεία. Τώρα, το κοινωνικό ταμείο, εδώ πέρα τα ποσοστά πληρωμών είναι υψηλότερα. Είναι πιο εύκολο να δοθούν, αν θέλετε, οι πόροι αυτοί. Το ίδιο και στο Ταμείο Συνοχής. 14% ποσοστό πληρωμών, 14,2%. Ωστόσο, το 66% των κρατών βρίσκονται κάτω από το επίπεδο αυτό και ορισμένες χώρες βρίσκονται στο 7%. Και πάλι η κατάσταση εδώ πέρα δεν είναι ίδια με άλλα ταμεία. Για παράδειγμα, στο κοινωνικό ταμείο, στα soft loans, οι χώρες με, το, με τις μεγαλύτερες πληρωμές από το κοινωνικό ταμείο έχουν τα χαμηλότερα requirement rates, τα μικρότερα ποσοστά απαιτήσεων. Και υπάρχουν και χώρες που είχαν δυόμιση φορές περισσότερα χρήματα που δόθηκαν κατά κεφαλή και για τις οποίες το ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν χαμηλό, 2%. Αν πάτε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εδώ πέρα το μέσο ποσοστό που έχουμε απαιτήσει είναι 9,3%, κάτω δηλαδή από το κοινωνικό ταμείο και το 56% των χωρών βρίσκονται κάτω από το επίπεδο αυτό. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν acquirement rate της τάξης του 4,5%. Επομένω, αν δούμε το Ταμείο Συνοχής που απευθύνεται σε 15 χώρες μέλη, όχι σε 27, σε 15 χώρες μέλη μόνο που απευθύνεται το Ταμείο Συνοχής, βλέπουμε ότι το fulfillment rate είναι 12% και 60% βρίσκονται κάτω, το χώρο βρίσκονται κάτω από το 10% και το χειρότερο ποσοστό fulfillment είναι 6%. Και γι' αυτό το λόγο είπα στην συγγήτρια την συντονία ότι δεν αρκεί να λέμε ότι βελτιώνεται η εφαρμογή ορισμένων προγραμμάτων. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε σαν συμπέρασμα της κατάστασης είναι να δούμε τι γινόταν την περίοδο 2000 με 2006. Τέσσερα δισεκατομμύρια δεν απορροφήθηκαν και αν παραμείνει το ποσοστό απορρόφησης στο ποσό, στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, σίγουρα τα πράγματα θα επιδεινωθούν στο μέλλον. Αυτό για όλα τα ταμεία, και για το Ταμείο Συνοχής και για το Κοινωνικό Ταμείο. Για ορισμένα από τα ταμεία αυτά χρειάζεται να δοθεί και μια περίοδος παράτασης. Σας τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιούνται, οι πόροι δεν θα απορροφούνται και τότε η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αυτούς για άλλες ανάγκες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν δοθούν τα χρήματα αυτά σε κάποιες άλλες ανάγκες, σίγουρα θα απουσιάσουν από τις ανάγκες που υπάρχουν στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής. Τώρα όσον αφορά την ε, γνωμοδότησή μου, Βλέπουμε κάποια θετικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο τέλος του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την συμπερέλαβε στον προπολογισμό προκειμένου να αυξηθούν οι προκαταβολές για το Ταμείο Συνοχής και δόθηκαν οι προκαταβολές αυτές με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πληρωμές. Ουσιαστικά όμω το αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, δεν είναι πάρα πολύ ψηλό. Φτάσαμε μόνο σε ποσοστό 8%. Οι επόμενε όμως, οι επόμενες προτάσεις που γίνανε ήταν οι εξή. Αρχικά μια πρόταση του Ιουλίου του 2009 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε οι χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση να μην συγχρηματοδοτήσουν τα κοινωνικά ταμεία και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάμβανε εξ ολοκλήρου την χρηματοδότηση αυτή. Γίνανε απαραίτητοι υπολογισμοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φτάσανε στα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δούμε τον προπολογισμό του 2010, η διαφορά ανάμεσα στις ε, πληρωμές και την ανάληψη υποχρεώσεων είναι 2,5%. Από ό,τι γνωρίζω όμως, αν δείτε την συσσωρευμένη διαφορά ανάμεσα στις πληρωμές και τις υποχρεώσεις από το 2007 και μετά, στο κοινωνικό ταμείο η διαφορά είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ και πληρωμές 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφορά της τάξης των τριών περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σύστημα αυτό των, της προκαταβολής κάποιων πληρωμών προτάθηκε κυρίως από το Συμβούλιο, αφού είναι εμφανές, και αν δώσει κανείς σημαντικές προκαταβολές στην αρχή, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο τέλος της δημοσιονομικής περίοδου. Και λοιπόν, για αυτό το λόγο, το Συμβούλιο αρνήθηκε να γίνει κάτι τέτοιο και γι' αυτό είπαμε κι εμείς με τους υπόλοιπους συγητήσεις ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση αυτή. Καταρχά δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι στον τρέχοντα προπολογισμό στα ταμεία αυτά. Δεν πρέπει να πάρουμε πόρους από τα υπόλοιπα ταμεία για να κάνουμε τις προκαταβολές αυτές. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιτρέπει στις εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν κάτι τέτοιο. Και έπειτα είπαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν θα ήταν σε θέση να συγχρονοτοδοτήσουν σε αυτό το επίπεδο για να συμβάλλουν. Το Συμβούλιο ενέκρινε μια διαφορετική απόφαση στη συνέχεια, την οποία ενέκρινε χθε η Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Οι πολιτικέ ομάδε αποφάσισαν να μην τροποποιήσουν την τελευταία αυτή πρόταση του Συμβουλίου. Τη σχολιάζω και την πρόταση αυτή στην έκθεσή μου. Το Συμβούλιο ουσιαστικά είπε ότι τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολλά, δεν μπορούν να πληρωθούν και γι' αυτό το λόγο μόνο ορισμένε χώρε στι οποίε έχει μειωθεί το ΑΕΠ του κατά 10% την περίοδο 2008-2009 και αυτές που έχουν άμεσες ε, Χρηματοδοτήσει άμεσα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι μόνε που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τι προκαταβολέ αυτέ. Καταλαβαίνετε ότι οι χώρε αυτέ βρίσκονται ουσιαστικά εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέντε είναι οι χώρε αυτέ, θα τι δείτε στο παράρτημα 1 και στο παράρτημα 2 θα δείτε ότι χρειάζονται 1,4 δισεκατομμύρια για τη συνοχή και 1,3 δισεκατομμύρια για το κοινωνικό ταμείο. και προσπάθησα να δω αν οι χώρες αυτές που βρίσκονται στο παράρτημα έχουν ε, τα απαραίτητα τα κατάλληλα acquirement rates. Για ποιο λόγο έχουν επιλεγεί αυτές και όχι κάποιες άλλες. Θα μπορούσα να πω ότι οι χώρες αυτές βρίσκονται σαστικά πάνω από τον μέσο να μέσα στις χειρότερες. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ε, μείωση του ΑΕΠ, ανάμεσα στο δημόσιο έλλειμμα των χωρών αυτών και των απαιτήσεων χρηματοδότησης. Από δημοσιονομικής πλευράς όμως τελευταία αυτή η πρόταση μπορεί να γίνει δεκτή, γιατί δεν απαιτούνται τόσα πολλά, τόσοι πολλοί πόροι, αλλά και από την άλλη θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο υπάρχουν τόσες μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Δεν μπορούμε να επικρίνουμε μόνο την Γενική Διεύθυνση περιφερειακή ανάπτυξη, ή γενικότερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές πέντε φορές περισσότερο, για παράδειγμα, στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας σε σχέση, μια σε σχέση με μια άλλη. Ε, εσωτερικά, στο εσωτερικό των χωρών το τοπίζονται συνήθως τα προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο στην γνωμοδότησή μου λέω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε, αν θέλετε, το σενάριο της ελάχιστης προσέγγισης. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τα τεράστια ποσά. Ζητάμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ένα διορθωτικό προπολογισμό για 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι για άλλα ποσά και λέμε επίσης στη συνέχεια ότι θέλουμε να δούμε ποια είναι η ανάληψη υποχρεώσεων που γίνεται. Ο κύριος Λαμασούρ θα πρέπει να γνωρίζει ότι πολλές φορές σε μηνιαία βάση πρέπει να υποβάλλονται διάφορες πληροφορίες και οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται στο ποσοστό πληρωμή σε σχέση με μια αρχική ανάληψη υποχρέωσης. Καταλήγεται λοιπόν σε κάποια ποσοστά τα οποία μπορείτε να δείτε και στο παράρτημα 1 και από την ε, μία πληρωμή στην άλλη, από τη μία ανάληψη υποχρέωση στην άλλη, οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν δεν είναι ε, αντιπροσωπευτικές. Πολλές φορές μπορούν να δώσουν μια ανθασμένη εικόνα. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να έχουμε κατά νου το εξής, κάτι που είναι πολύ σαφές. στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης του προπολογισμού, σε κάποιο ενδιάμεσο τέλο πάντων στάδιο, θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο τα ποσοστά μας είναι τόσο χαμηλά, για ποιο λόγο δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να δείτε και στην εκθεσή μου. Ευχαριστώ. Okay, merci, euh, Ευχαριστώ τον εισηγητή. αξιολογώτε η εισηγησή σας. Αξίζει νομίζω μια συζήτηση. Πολλοί ζήτησαν το λόγο. Προτείνω να μεταφέρουμε τη συζήτηση για την άλλη εβδομάδα. Θα βάλουμε και την προθεσμία για τις οπολογίες για μετά τις 4 Μαρτίου, ούτως ώστε να έχουμε μια καλή συζήτηση και να κυκλοφορήσουμε και τα παρατήματα με τα στοιχεία που μας έδειξε στον πίνακο ο κ. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η πνευματική του ικανότητα ήταν πολύ ψηλότερη από τις ικανότητες τις τεχνικές. Κάτι που είναι ένα θέμα βασικό αυτό, το οποίο δεν είχε απασχολήσει πολύ την Επιτροπή μας μέχρι τώρα και σίγουρα η Κομισιόν θα έχει πολλά να πει επ' αυτού. Υπενθυμίζω ότι στην Επιτροπή θα προβλέπεται η ψηφοφορία στις 16 Μαρτίου, άρα μπορεί να έχουμε προθεσμία για τις απολύγες λίγε μέρες νωρίτερα και θα παρουσιάσουμε την γνωμοδότησή μας προς την Περιφερειακή Επιτροπή, προς την Περιφερειακή Επιτροπή, συγγνώμη, που θα ψηφίσει στις 8 Ιουνίου. Ευχαριστώ τον κύριο Γκοντμάνης. Προτείνω να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του θέματος την άλλη εβδομάδα. Έτσι. θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο στην Έλγα Τρίπελ για να μας παρουσιάσει τις κατώντας ειδήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές του προπολογισμού του 2011 για τα λοιπά τμήματα. Καλωσορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα και τους συνεργάτες του που έφτασαν που θα καθίσουν στην ε, τιμόμενη θέση που παλιά είχε, προηγουμένως είχε ο πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έλγα, πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω με το κεντρικό στρατηγικό θέμα. Ξέρετε όλοι ότι μετά από μακρές ε, συζητήσεις υιοθετήσαμε επιτέλους τις συνθήκη της Λισαβόνας και για πρώτη φορά εργαζόμαστε βάσει των νέων κανόνων ε, προετοιμάζει του προπολογισμού για το επόμενο έτος. Αφενός έχουμε μια πολιτική προσέγγιση βάσει οποίας εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα θα πρέπει να είναι σε θέση μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων να αντιδράσουν στις νέες αρμοδιότητες που προσφέρει το συνδείξη της και που θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε. Δεν εξετάζουμε το θέμα αυτό για πρώτη φορά. Μα έχει απασχολήσει ήδη στα πλαίσια του προβλησμού 2010. Πολύ μεγαλύτερη όμω είναι η προσκλήση για τον προβλησμό 2011. Εγώ και μετά που θα ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Βέλε θα επανέλθω στο θέμα αλλά θα ήθελα να έχετε μια πρώτη ιδέα τι έχω κατά νου για τον προπολογισμό του 2011. Ναι, είναι σωστό. Οι δυνατότητες του Κοινοβουλίου μας και άλλων θεσμικών οργάνων μπορούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες της Λισαβόνας. Αυτό το 20% ε, που προέρχεται για τον προπορισμό του Κοινοβουλίου από το 1988 δεν είναι δεσμευτικό για μένα γιατί αν έχουμε τώρα μια νέα ε, συμβατική βάση, με μια διεύρυνση, με μια νέα ε, κατάσταση πολιτική από την οποία ανεκκινούμεθα, θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοστούμε. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε βέβαια στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης. Είναι προφανές ότι οι προπολογισμοί των κρατών μελών είναι πάρα πολύ περιορισμένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις απαιτήσει μας. Αλλά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και μια πολιτική μετριοπάθεια, αν θέλετε, όσον αφορά τις δυνατότητες του προπολογισμού μας σε σχέση και με τον προπολογισμό της Κομισιόν ή του, του Συμβουλίου. Αναφέρθηκε ένα στοιχείο 22%. Κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολικό αυτό. Χρειαζόμαστε πολλές συζητήσεις για το θέμα. Οπωσδήποτε και αυτό είναι σημαντικό και εδώ στο σώμα μεταξύ της Επιτροπής Προπολογισμών και του Προεδρείου και του Γενικού Γραμματέα βέβαια, αλλά και όσον αφορά την Κομισιόν και το Συμβούλιο, έχουν να πω ότι όταν υπήρχαν κάποιες συμφωνίες, ακόμα και αν είναι πολύ παλιές, όπως παραδείγματος χάνει Γενάρη 1988, ε, θα πρέπει να έχουμε συζητήσεις. ή συζητήσεις οι οποίες θα παρουσιάζουν τα συμφέροντα των εκάστοτε θεσμικών οργάνων, και τις δυνατότητες επικοινωνίας. Δεν επιτρέπεται να καταστρέψουμε τις άγουσες της επικοινωνίας. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό θέμα. Μπορούμε να δεχτώ να κινηθούμε κάπως, αλλά κατά γνώμη υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια που θα πρέπει να τα εξετάσουμε πολιτικά και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πολιτικά ευφυώς για να μην υπερβάλλουμε σε καμία στιγμή. Αυτή τη στιγμή η έκθεση που σας υποβάλλω αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση. Πολλά θα πρέπει να διευκρινιστούν τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, δεν θέλω να προτρέξω των εξελίξεων. Εγώ θέλησα να αναφερθώ σε κάποιες σκέψεις. Καταρχήν το θέμα της, ε, του αποδεκτού οικολογικά των κτίριων μας και τι μπορούμε να αλλάξουμε. Είναι ένα θέμα με τα αυτοκίνητα, τι θα γίνει με το λεγόμενο job ticket για τους απασχολούμενους. Μετά ε, εξετάσουμε και το θέμα όσον αφορά το καθεστώς Microsoft εδώ στο σώμα. Sollten wir auch hier im Hause äh, unsere Öffnungsregeln dem Υπάρχουν πολλά που θα μπορούμε σωστά ίσως να αλλάξουμε. Για διαδικασία, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν καλό να ακούσουμε τώρα τον Γραμματέα, τον κύριο Βέλε, και ίσως θα μπορούσα να πάρω το λόγο μετά για, και να αναφερθώ στο τέλος και στα σχόλια του συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κάτι μόνο που είπε η Έλγα, την οικολογική συμβατότητα του κτίριου. Να σας πω στους συναδέλφους ότι στη Γαλλία Ξεκινήσαμε ένα ε, πλαίσιο εξαιρετικής αποτελεσματικότητας που ενθαρρύνει την κάλυψη των σκεπών των δημοσίων κτηρίων με φωτοβολταϊκά πάνελ. Ο ηλεκτρισμός που παράγεται με τον τρόπο αυτό αγοράζεται από τον βασικό από την ε, βασική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην EDF, σε τιμή 20 φορές ακριβότερη από την ε, τιμή αγοράς. Τρελή δηλαδή ε, η εξαιρετική ε, αποτελεσματικότητα, απαράδεκτη, απαράδεκτο κόστος κάπως. Θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τα δύο. Αυτό το λέω για τους Βέλγους φίλους, μπορούν να βρουν ενδιαφέρουσα την ιδέα για τη χρησιμοποίηση στα κτίρια του Κοινοβουλίου που βρίσκονται στο Βέλγιο. Ο κανόνα αυτό θα εφαρμοστεί και για τα κτίρια του Κοινοβουλίου που βρίσκονται στο Στρασβούργο και να αποτελέσουν σχολείο για τα κτίρια του Λουξεμβούργου. Κύριε Γενική Γραμματεύ, θέλετε να μιλήσετε τώρα, στο τέλος, παρακαλώ. λύστε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Συγγήτρια αξιότιμοι βουλευτέ. Σα ευχαριστώ για την δυνατότητα που έχω να ενισχύσω την συζήτηση για τις κατευθύνες γραμμέ. Το Προεδρείο το συζήτησε σε ένα πρώτο γύρο και αύριο στην συνεδρίαση του Προεδρείου πρόκειται να απόφαση. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο βέβαια σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτή τη στιγμή. Στις 8 Μαρτίου θα εξετάσουμε τα προκαταρτικά ε, στοιχεία και στις 24 Μαρτίου, εάν υπάρχει πολιτική υποστήριξη, θα καταλήξουμε ενδεχομένω σε μία απόφαση. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια ε, σχετικά με αυτά που είπε ιδίως για τη Λισαβόνα. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα προκοδοτηθεί το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε τα δικαιώματά μας στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας να μην παραμείνουν κενό γράμμα, αλλά να μπορέσουν να προεκτελεστούν. Πρόσφατα είχα τη δυνατότητα να συζητήσω με έναν ε, υφυπουργό από τη Γερμανία που μου είπε ότι στο Υπουργείο του 200 υπάλληλοι ε, συνεργάζονται τακτικά σε ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Αν σκεφτούμε πόσο, ε, ποιο είναι το συλλογικό know-how, το τεχνογνωσία όλων των ανθρώπων αυτών, πραγματικά θα πρέπει να έχουμε και εμείς ανάλογες ε, γνώσεις για να μπορούσαμε να είμαστε ισότιμοι νομοθέτες. Και γι' αυτό τα επόμενα χρόνια θα πρέπει ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου να εστιαστεί στην πολιτική ενίσχυση των βουλευτών. Το πρώτο βήμα θα είναι ο συμπληρωματικός προπολογισμό ε, για το 2010 με η ψηφοαναλυτική υποστήριξη για τις ε, επιτροπέ τις ε, πολιτικές ομάδες και τις γραμματείες των μεμονωμένων βουλευτών και κατόπιν προβλέπεται και η έμεση υποστήριξη των βουλευτών μέσω του ε, τμήματος πολιτικής υπάρχει ένα policy department για τον προπολογισμό και θέματα προπολογισμού που βοηθάει τους βουλευτές και επίσης και μέσω της βιβλιοθήκης μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και θα μπορούμε να έχουμε και, και στην πραγματική υποστήριξη. Βέβαια προβλέπεται πέρα από το διευθυντικό προπολογισμό του 2010 να υπάρχει και ένα δεύτερο τμήμα των ισχύσεων της γραμματείας ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα και συμπληρωματικού συνεργάτη για τους βουλευτές. Πέραν αυτών υπάρχουν και διάφορες ε, θεσμικές υποχρεώσεις. Ακόμα και δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει με το Συμβούλιο, ποιος θα είναι ο μηχανισμός για την ε, επιλογή των συμπληρωματικών 18 βουλευτών βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, συμφωνούμε ότι θα υπάρξουν 18 επιπλέον βουλευτές. Οι βουλευτές αυτοί, κατά πάσα πιθανότητα, θα αναλάβουμε τι εργασίε εδώ στο Κοινοβούλιο το 2011. Γιατί η εκλογή των συμπληρωματικών αυτών βουλευτών προϋποθέτει σε πολλές χώρες τροποποίηση του πρωτογενούς δικαίου και θα πρέπει να υπολογίσουμε μία περίοδο επικύρωσης ενός έτους. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να προβλέψουμε τους πόρους για να μπορέσουμε να προκοδητήσουμε αυτούς τους συμπληρωματικούς βουλευτές για να μπορέσουν να ασκούν το αξιωμά τους, γιατί θα είναι πλήρης βουλευτές. Δεύτερο, η διεύθυνση προς την Κροατία είναι όσο πάει και πιο πιθανή. Αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα και από τις πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων ετών. Θα υπάρξουν συμπληρωματικά κεφάλαια. Εμείς θεωρούμε ότι αρχές του 2012 θα υπάρχουν ενδεχομένως Κροάτες βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι ήδη το 2011 θα πρέπει να αρχίσουμε, οι δύο γλωσσικές υπηρεσίες, να δημιουργούμε ε, δυναμικό και για την κροατική γλώσσα. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την πλήρη υπογλωσία και για τους Κροάτες βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι παραδοσιακά προβλέπονται 124 θέσεις συνεργαστών για τις χώρες διεύρυνσης. Αυτή τη στιγμή η μισή περίπου θα προβλεφθούν ήδη το 2011 για Κροάτες συνεργάτες, αλλά κυρίως όσον αφορά τις γλωσσικές υπηρεσίες. Στην πρώτη φάση, εφόσον δεν έχει ε, επικυρωθεί η συνθήκη, με κάποιες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Είναι επίσης παράδοση του σώματος εδώ. Ε, λίγο καιρό πριν έχουμε παρατηρητές από τις χώρες αυτές υποψήφια μέλη. Γι' αυτό το έτος 2011 θα πρέπει να προβλέψουμε πόρους για να μπορέσουμε δυνατότητα παρατηρητές από την Κροατία να συμμετέχουν στην εργασία του Κοινοβουλίου. Υπάρχει και ένα τέταρτο θέμα, είναι τα απολετή προγράμματα. Στο περσινό προπολογισμό κάναμε καταρχήν την εισαγωγή σε ένα τριετές ε, πρόγραμμα για τα κτίρια, που ξέρετε ότι μετά από κάποια προβλήματα οδηγηθήκαμε στην ανάγκη αυτή και γνωρίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω και να έχουμε και ίδιο δυναμικό για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τις εργασίες των εξωτερικών εμπειρογνωμών. Για το 2011 θα ήταν το δεύτερο έτος του τρίτου αυτού προγράμματος. Θα ήθελα να σας πω και είναι σημαντικό νομίζω ότι κατόπιν πρόσκλησης του σε επιτροπές προπολογισμών αυτές το Προεδρείο έχει προχωρήσει σε μια μέσο και μακροπρόθεσμη πολιτική για τα κτίρια. Το Προεδρείο δημιουργήσε μια ομάδα εργασία και νομίζω ότι θα ικανοποιήσει αυτό την κυρία Τρίπελ. Μια ομάδα εργασία λέω που δεν ασχολείται μόνο με κτίρια, αλλά κτίρια, μεταφορές και το λεγόμενο πράσινο κοινοβούλιο προσπαθεί να εξετάσει οικολογικά θέματα, θέματα μεταφορών και ταυτόχρονα τα θέματα των κτηρίων. Γιατί τα τρία αυτά θέματα δεν μπορούμε λογικά να τα αποχωρήσουμε. Η ομάδα εργασίας αυτή έχει προχωρήσει πολύ και θεωρώ ότι η σβάθο συζήτηση για μια μακροπρόθεσμη προληπτική κτηρίων θα γίνει στο Προεδρείο στις 8 Μαρτίου και κατά πάση μετά η απόφαση στις 24 Μαρτίου, ούτως ώστε τα αποτελέσματα της ε, πολιτικής αυτής για τα κτίρια θα μπορέσει να ληφθεί υπόψη επαρκώ στην διαδικασία για τον προπολισμό του 2011. Καταρχήν θα πρέπει να συμφωνηθούν κριτήρια για την κάλυψη του χώρου, ποιος θα πρέπει δηλαδή να δικαιούται πόσο χώρο και για ποιους λόγους. Αυτό δεν έχει ε, ενημερωθεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι υπάρχουσε επιφάνειε, ποιε είναι οι ενδεχόμενε συμπληρωματικέ επιφάνειε που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε έτσι μια πολιτετή στρατηγική. Το ίδιο ισχύει στον τομέα τη πληροφορική και εκεί στα πλαίσια τη περσινή διαδικασία για τον προεπορισμό είχε κληθεί το Προεδρείο να προετοιμάσει μια μέσο και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον τομέα η ομάδα εργασία έχει αρκετά προχωρήσει ήδη και ελπίζω ότι πραγματικά τέλη Μαρτίου θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε στο Προεδρείο και για το θέμα της πληροφορικής και στρατηγικής ICT. Σημαντικό είναι επίση να υπάρχει καλή εξορρόπηση μεταξύ εσωτερικόποίηση και εξωτερικοποίηση, γιατί αυτή τη στιγμή πολλοί τομεί εξαρτώνται από εξωτερικούς ε, προσφέρει στις υπηρεσίες και δεν έχουμε κανένα επαρκή έλεγχο για την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάπως περισσότερες εσωτερικές ε, δυνατότητες, εσωτερικό δυναμικό, για να μπορέσουμε να ελέγχουμε και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Εκ έχουμε τον τομέα των γλωσσικών υπηρεσιών, και αυτό ήταν πάρα πολύ στα πλαίσια της Μάκα. και εδώ θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κατά το μέγιστο τους πόρους που προβλέπονται. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι γίνεται ήδη σωστή κατανομή μεταξύ των διαφόρων γλωσσών. Θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε σε μια κατανομή βάσει των πραγματικών αναγκών, όχι των υποθετικών αναγκών που είχαμε λάβει υπόψη από πέντε χρόνια. Υπάρχει και ένας ειδικό παράγοντος, σημαντικός Όπω ξέρετε το Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε με το Βέλγιο σε σχέση με την ε, νέα, με την κατασκευή συγγνώμη, νέων κτηρίων και τον εξοπλισμό του. Τώρα έχει το Κοινοβούλιο λάβει 86 εκατομμύρια περίπου και τίθεται το θέμα της χρησιμοποίησης τους. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλό το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά μακροπρόθεσμα σαν επένδυση και να μην τα χρησιμοποιήσει στην καθημερινή εργασία. Τώρα, ποια θα είναι η πραγματικά σωστή επένδυση θα πρέπει να το σκεφτούμε. Αλλά οπωσδήποτε εδώ έχουμε ξαφνικά λάβει ένα ποσό που αξίζει να μελετήσουμε πώς θα το χρησιμοποιούμε σωστά και προς όφελος του Κοινοβουλίου μακροπρόθεσμα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τον πολύ καλό διάλογο που είχα μέχρι τούδε με την κυρία Τρίπελ. Όπως σας είπα, εδώ πρόκειται για πρώτες καταρχήν συζητήσεις. Αριθμικά στοιχεία θα υποβληθούν στο Προεδρείο στις 8 Μαρτίου και οι ενδεχομένω θα ε, αποφασιστούν, θα ψηφιστούν στις 24 Μαρτίου με τις ενδεχόμενες τροπολογίες. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα. Πάρα πολύ πλήρη η παρουσίασή σα και πάρα πολύ σαφή. Πολλοί έχουν ζητήσει τώρα το λόγο. Έχουμε κάπου 20 λεπτά. Προσπαθώ να είμαι σύντομη λοιπόν. Ο κύριο Φόβελ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να υποστηρίξω την ε, έκθεση συγγήτριας. Σίγουρα το όλο εγχείρημα θα ήταν ε, πολύ δύσκολο γιατί δεν ε, είχαμε λάβει τις κατευθυντήρες γραμμές από το Προεδρείο. Πράγμα το οποίο έκανε και τη δουλειά των ίδιων των συναδέλφων πολύ δύσκολη καθότι έπρεπε μέχρι την Πέμπτη να υποβληθούν οι τροπολογίες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα. Το κατόφλι του 20% όπως και η συγγήτρια, έτσι και εγώ καταλαβαίνω ότι η διάσκεψη των Πρόεδρων προτείνει εδώ πέρα μια αύξηση του κατοφλίου αυτού από το 20% στο 22%. Παρουσία σας έγινε αυτό το πράγμα κύριε Πρόεδρε. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη κύριε Πρόεδρε ζητάνε από το Προεδρείο να συνεργαστεί μαζί μας προκειμένου να συμφωνηθεί το 22% ή μας ζητούν να βρούμε ε, τρόπους χρηματοδότησης αφού το 22%. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας δώσετε και τη δική σας γνώμη του ζητήματος. Και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία ενδεχομένω θα πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή μας είναι τα ενσωματωμένα συστήματα διαχείρισης της γνώσης, τα μέλη έχουν τους διαθέσιμους πόρους και νομίζω ότι θα πρέπει να τους χρησιμοποιούν είτε πρόκειται για το παρατηρητήριο, είτε πρόκειται για τους, ο, τις δυνατότητες που δίνονται μέσω διαδικτύου, είτε τα ψηφιακά μέσα. Επίσης, το ζήτημα της πολιτικής για τα κτίρια, της στρατηγικής για τα κτίρια. Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να ολοκληρώσουμε τη στρατηγική αυτή, να υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση, να ξέρουμε και ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσει και ενδεχομένω να συνεργαστούμε και με άλλα θεσμικά όργανα. Ενδεχομένω να μοιραζόμαστε με άλλα θεσμικά όργανα κτίρια, όπω μοιραζόμαστε γνώσει ή κόστο πολλέ φορέ. Επίση, το προσωπικό που θα πρέπει να πάει προς την γραμματεία της Επιτροπής μετά την έναρξη της ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνα το προσωπικό δίδεται προς τις επιτροπές, με βάση το βάρος εργασίας που έχουν, το βάση το άχθος εργασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε πάνω κάτω ποιο θα είναι αυτό το άκθος του 2011 προκειμένου να γίνει η απαραίτητη κατανομή. Ενδεχομένως θα πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο και το ζήτημα της, του καναλιού Europarla TV να δούμε αν ε, ο υφιστάμενος τρόπος διαχείρισης του καναλιού αυτού είναι ο καλύτερος και έπειτα να δούμε τις σταθερές μας δαπάνες, όπως για παράδειγμα η μισθή, αλλά και τις ε, δαπάνες που παρουσιάζουν κάποια διακύμανση. Ενδεχομένως αυτές θα πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα στο μέλλον. Αυτά πιστεύω ότι είναι τα σημαντικότερα ζητήματα, οι βασικότερες προτεραιότητες και νομίζω θα υποβληθούν και κάποιες τροπολογίες σχετικά. Ο κύριος Φέρναντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον εισηγητή μας, την εισηγήτρια, για την εξαιρετική εργασία και ευχαριστώ και τον Γενικό Γραμματέα που ήρθε στην Επιτροπή μας σήμερα. Κατανοώ τις προτεραιότητες που ανέθεσε την νομοθετική δραστηριότητα και εγώ πιστεύω ότι τα μέτρα που προβλέπονται για βουλευτές, ομάδες και επιτροπές είναι σωστά και σκόπιμα. Πιστεύω ότι η κατάσταση έχει ως εξής. Έχουμε έναν προϋπολογισμό επί του οποίου συμφωνούμε. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε τους πόρους αυτούς. Εάν αποσύρουμε 126 εκατομμύρια για τα προγράμματα ανοικοδόμησης, προφανώς τα χρήματα αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα για άλλη δραστηριότητα. Αυτό είναι προφανές. Αυτό που θεωρώ σημαντικό λοιπόν είναι να δούμε ποιο είναι το τμήμα των υποχρεωτικών παγίων δαπανών και να δούμε τα όρια που είναι αναγκαία για να γίνει μια σωστή νομοθετική δραστηριότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα πρέπει να δούμε το ποσό, το μήνυμο ποσό που χρειάζεται για να υπάρξει μια σωστή νομοθετική δραστηριότητα, πώς να επιβιώσουμε με μια σωστή αξιοπρεπή δουλειά. Τι χρειαζόμαστε, 20-22%? Αυτό εξαρτάται από μια σειρά στοιχείων. η κατηγορία 5 θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διοικητικές δαπάνες κατά την άποψή μας. Το 20% ίσως να μην να είναι πολύ. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι σταθερές δαπάνες, οι πάγιες δαπάνες, οι υποχρεωτικές δαπάνες και κατόπιν να ορίσουμε κάποιος, κάποια κριτήρια στον τομέα της σωστής διάφανης διαχείρισης. Τέλος, δε, να δούμε τι χρειαζόμαστε. Βρισκόμαστε ακόμα σε μια πειραματική φάση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να δείξουμε μια κάποια ευελιξία, να ορίσουμε κάποιες θέσεις, να δούμε τι χρειάζεται μετά, να κάνουμε μία δουλειά που να περιλαμβάνει στοιχεία διαφάνειας, αλλά και βιωσιμότητα. Αυτό αφορά μια σειρά κατηγοριών, την πολιτική ακινήτων π.χ. Να μην μπούμε σε αγορές που θα εξαντλήσουν γρήγορα τον προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τη διάρκεια θα πρέπει να ξέρουμε πού βαρίζουμε. Και νομίζω ότι από αυτού συμφωνούμε όλοι. Δείτε για παράδειγμα αυτή την ερμηνεία του 20%. Εγώ συμφωνώ ότι επιβάλλουμε κάποια όρια στους εαυτούς μας. Σωστό. Λογικό. Και εμφανίζεται και στο σχέδιο ψηφίσματος για τον διοθωτικό προπολογισμό. Συμφωνούμε, έλεγα, εμπολής με το περιεχόμενο της, έκθεση, της έκθεσης. Ίσως να πρέπει να δούμε κάπως καλύτερα το θέμα της μετάφρασης. Μας λέει, η έκθεση λέει ότι πρέπει να είναι με επαρκή προσόντα, qualified. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Μετά, γίνεται λόγος για τις μη διακρίσεις. Και αυτό το πράγμα είναι λίγο ασκατανόητο. Το κείμενο δεν ε, ξεκαθαρίζει. Υπάρχουν διακρίσεις, γιατί ζητάμε να υπάρχουν μέτρα κατά των διακρίσεων. Μήπως η συγγήτρια μπορούσε να μου δώσει κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις. Αυτά. Αυτά. Επαναλαμβάνω. Να γνωρίζουμε ποιες είναι οι σταθερές υποχρεωτικές, οι πάγιες υποχρεωτικές δαπάνες μας, πρώτο πράγμα, και κατόπιν να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Είτε τηρούμε το 20% και αν μείνουμε κάτω από το 20% στο καλύτερο, αλλά να δούμε τέλος πάντων πού βρισκόμαστε. Υπάρχουν ορισμένες μεταβλητές δαπάνες, αλλά πάντα πρέπει να δούμε τη σχέση κόστους όφελους και πάνω στη βάση αυτή θα πρέπει να λάβουμε την τελική μας απόφαση. Πιστεύω ότι αν κάνουμε αν προχωρήσουμε έτσι, θα έχουμε την υποστήριξη όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η νομοθετική δραστηριότητα είναι μια σημαντική δουλειά, κοστίζει, είναι δαπανηρή, δεν γίνεται τζάπα και πρέπει να νομοθετήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Έχω πολλούς που έχουν ζητήσει το λόγο να είστε πάρα πολύ σύντομοι γιατί μόνο 10 λεπτά έχουμε. Ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για το 20%. Χρειαζόμαστε μια νέα φόρμουλα για το μέλλον. Ε, ο κανόνας αυτός έχει, είναι, είναι 20 χρονών. Αν δεν υπήρχε η συνθήκη της Λισαβόνας και το καθεστώς των μελών, δεν θα μιλούσαμε για τη φόρμουλα αυτή. Και νομίζω ότι τούτο μας δίνει και μια εικόνα προς τα πού θα πρέπει να πάει το νούμερο αυτό, πώ πια κατεύθυνση να στραφεί. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα που αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες. Πριν από ένα χρόνο τα μέλη του Κοινοβουλίου έστειλαν ένα σαφές μήνυμα. Όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου το 2010 θα πρέπει να είχαν τη δυνατότητα να ασκούν τις δραστηριότητες σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν. Χαίρο που το Κοινοβούλιο προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση αυτή και ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα για τις δραστηριότητε του προ την κατεύθυνση αυτή. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα κείμενά μα. Πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό σχέδιο στο Κοινοβούλιο που λεγόταν Interpretation ad personam. Πέρσι ήταν η πρώτη, ε, τέτοι, η πρώτη χρονιά χρήση ενός τέτοιου, μιας τέτοιας δυνατότητας. Είχαμε μια κατανάλωση 100.000 ενώ ο προπολογισμό ήταν 4 εκατομμύρια. Ελπίζω του χρόνου αυτό να είναι υψηλότερο το ποσοστό φέτος. Για τις γλώσσες, το ελεκτικό συνέδριο είπε ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης και εξοικονόμησης όχι μόνο στο Κοινοβούλιο αλλά σε όλα τα όργανα. Γι' αυτό το 2010 υιοθετήσαμε μια οριζόντια πρόταση που έθεσε στο αποθεματικό για όλα τα θεσμικά όργανα 5% εξωτερικών μεταφράσεων. Αυτό θα πρέπει να το συνεχίσουμε και το 2011 βλέποντας τι συνέπειες έχει και πώς να προχωρήσουμε για το μέλλον. Όλα τα έτη, όλα τα ο φέτος περιμένω όλα τα ε, θεσμικά όργανα να εξετάσουν την τηλεεργασία των μεταφραστών και να κοιτάξουν όλα τα όργανα να δουν τι, τι συνέπειες οικονομικές έχει κάτι τέτοιο. Θέλω να δούμε και θα ζητήσουμε από όλα τα κράτη να δώσουν, ε, ε, όλα τα όργανα να δώσουν πληροφορίες για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μη ε, χρησιμοποιούμενες δυνατότητές τους από ανθρωποόρες μέχρι χώρο. Να, μην, να σας θυμίσω και την Συμφωνία Συνδιαλλαγής του Οκτωβρίου. Φέτος στο Κοινοβούλιο θα υπάρξει μια οργανωτική, ένας οργανωτικός έλεγχος στην Γενική Διεύθυνση και τις εσωτερικές υπηρεσίες. Αυτό θα δώσει πληροφορίες για, τις, ε, για την κατάσταση στο μέλλον. Πέρσι εγκρίναμε ένα κείμενο για το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας που δεν εμπλέκει τη δική μας ε, μόνο επιτροπή αλλά και άλλες. Επίσης, επισκέφθηκα το κέντρο επισκεπτών και είδα ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου επισκεπτών είχε στοιχεία, πληροφορίε, ε, όχι μόνο για την ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και την ιστορία του, ε, ε, για την ιστορία ε, της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας τους δουν μεταξύ τους λοιπόν ε, οι αρχιτέκτονες. Ο κύριος Πόρτας. Πρώτον, 20-22%. Δεν έχουμε απάντηση προς το παρόν. Δεν χρειάζεται να λάβουμε θέση. αν ακολουθήσουμε την πρόταση του ΕΡΚ, όλες οι διοικητικές δαπάνες να είναι στην κατηγορία 5, πρέπει να κάνουμε έναν υπολογισμό, να δούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Έχουμε από τη μία μεριά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και από την άλλη την εκτέλεσή του. Το ένα δεν είναι συναφές με το άλλο. η κατάσταση του Κοινοβούλου είναι διαφορετική από των άλλων οργάνων. Ναι, για συγκεκριμένους λόγους. Πρέπει να υπάρχει χωριστή εκμετάλλευση, χωριστή διαχείριση κάθε προπολογισμού. Τρίτο, τρίτη παρατήρηση. θα δαπανίσουμε πολλά χρήματα στην σωστή νομοθεσία για να έχουμε υποδομές, νέους υπαλλήλους κλπ. Θα δώσουμε λοιπόν πολλά λεφτά για να έχουμε μια καλύτερη δουλειά στον τομέα της νομοθετικής δραστηριότητα. Αν ωστόσο ταυτόχρονα δεν προχωρήσουμε σε μια ανάλυση δαπανών που είναι δικαιολογημένες ή όχι, τότε δεν προχωράμε σωστά. Αν δεν κοιτάξουμε ποιες δαπάνες είναι δικαιολογημένε, ποιες δεν είναι και αν δεν δούμε βουλευτές οι, οποίες παίρνουν, ε, βουλευτές οι οποίοι παίρνουν ε, μια σειρά αποζημιώσεων, να τα ταξί από εδώ, να τα ταξί από εκεί, είναι... Ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν δεν ξεκινήσουμε δηλαδή από το μηδέν για να δούμε τι δικαιολογείται και τι δεν δικαιολογείται, τι παίρνουμε και τι δεν πρέπει να παίρνουμε, ε, δεν θα έχουμε μια σωστή προσέγγιση. Τα ταξίδια. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν προτάσεις της Επιτροπής μέχρι τον Ιούνιο, γιατί γίνεται μια μελέτη σχετικά. Υπάρχουν μια σειρά μεταβλητών δαπανών. Αν δεν το δούμε από την αρχή, νομίζω ότι διασπαθίζουμε χωρίς λόγο τα έξοδά μας. Ο κύριος Φέρν. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ τη Χέλγα και τον κύριο Βέλε για, την παρουσία, για τις παρουσιάσεις τους. Έχω μία ερώτηση. Μιλούσατε συνεχώς για ανάγκη αυξήσεων. Συμφωνώ. Αλλά εμείς είμαστε επιτροπή προπολογισμών και άρα πρέπει να εξοικονομούμε για κάτι. Μπορεί ο Γενικό Γραμματέα να μα πει ποιε είναι οι προτεραιότητέ του για να υπάρξει εξοικονόμηση, εξορθολογισμό, κριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων δαπανών, αποτελεσματικότητα των λύσεων για τη μείωση του κόστου. Γιατί φαντάζομαι ότι και αυτό θα είναι κομμάτι των εκτιμήσεών σα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Πολλοί άλλοι έχουν ζητήσει το λόγο. Δυστυχώ, ωστόσο, δεν έχουμε χρόνο. Προτείνω να Μα στείλει γραπτό τι απαντήσεις του κύριος Γενικό Γραμματέας για τα ερωτήματα που του τέθηκαν και τον αφορούν ε, ευθέω και να δώσω το λόγο στην Έλγα για να κλείσει. Ζήτω συγγνώμη από του υπόλοιπου συναδέλφου. Έλγα, Θέλει να μας πεις τι συμπέρασματα καταλήγει από την ανταλλαγή αυτή απόψε. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά προτάσει βελτίωση, καλύτερη διαχείριση, καλύτερη οργάνωση που οδηγούν σε εξοικονομήσει, είμαι ανοιχτή. Βέβαια, από την άλλη μεριά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολιτική κατάσταση, σύμφωνα με οποία η δυνατότητα εργασία μα ε, και ημών και των επιτροπών μα ε, θέλουμε να βελτιωθεί. Αυτό είναι ο στόχο που δεν με βρήκε σύμφωνο, γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα στοιχεία, παρά μπορούμε να συζητήσουμε μόνο πολύ γενικά. Άμα προβλέψουμε τις προ... προβλέψεις ένα στοιχείο, αυτή τη στιγμή προβλέπεται ένα ε, περιθώριο για το 2009 109 εκατομμυρίων. Αλλά αυτά τα μέτρα ε, προβλέπουν συμπληρωματικά 160 εκατομμύρια συμπληρωματικά. Δηλαδή κατά πώ θα ανεβούμε στο 22% δεν καλύπτεται από το περιθώριο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αδέλφους για τις τοποθετήσεις τους. Θα προσπαθήσω τις επόμενες μέρες και όσον αφορά την πολιτική μου προσέγγιση και όσον αφορά συγκεκριμένε προτάσει, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μα. Ένα παράδειγμα. Δεν έχουμε πουθενά, παραδείγματο χάρη, είναι γραφή μπράγια για του τυφλού. Δεν είμαστε δηλαδή πολύ φιλικοί προ τα άτομα με δικές ανάγκε. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν θέλω να το αναπτύξω, αλλά σας λέω ότι θα θέλω να υποβάλω κάποιες προτάσεις και γενικά αλλά και συγκεκριμένες για βελτιώσεις. Ευχαριστώ. Très bien, je vous remercie. Donc, je vous propose rester là sur ce... Πολύ ωραία. Ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό. Το ζήτημα του κυρίου Άλβαρο θα πάει στην επόμενη συνάντηση γιατί ήδη έχουμε φτάσει στις 6.30 και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε άλλο τους δερμηνείς. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ Αέλγα, σας ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα στις 4 Μαρτίου στην επόμενη μας συνεδρία.